Buongiorno, colleghi, Συνάδελφοι, αρχίζουμε τις εργασίες μας, τις ακρόασεις στην Επιτροπή ΚΡΙΜ. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα σας πρότεινα να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 7ης και 27ης Μαΐου. Υπάρχουν αντιρρήσεις, φαίνεται πως όχι. Άρα θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά σας υπενθυμίζω ότι η συνεδρίαση αυτή ε, ακούγεται σε απευθείας αναμετάδοση μέσω της ιστοσελίδας μας και αργότερα προβλέπεται μία συνάντηση των συντονιστών από τις 4.30 και μετά στην ίδια αίθουσα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των πολιτικών προοπτικών. Στα πλαίσια αυτού του κλάστερ θα ακούσουμε τα δεδομένα από τις ε, μελέτες σε σχέση με τις ε, δημόσιες προμήθειες και την κατανομή των ε, κονδυλίων, των κοινοτικών κονδυλίων. Θα ακούσουμε τον Μάικ Μπέκ και Φρανσίσο Καρντόνα που θα μας μιλήσουν για τις πρώτες ε, εκθέσεις, τα πρώτα δεδομένα. Η συζήτηση θα έχει αυτή τη διάρθρωση. 15 λεπτά έχει στη διάθεσή του κάθε εισηγητής για να παρουσιάσει την ε, εισήγησή του. Μετά θα γίνει μία συζήτηση δίνοντας ε, προτεραιότητα στους συντονιστές. Δίνω το λόγο στους κυρίους, στον κύριο Μπέκ καταρχήν και μετά ο κύριος Καρδόνα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να παρουσιάσουμε τα προσωρινά μας αυτά συμπεράσματα. Λέγομαι Μπέκ και εργάζομαι στην Ουαδαλαχάρα της Ισπανίας, στην εταιρεία Mayer Sons, μαζί με τον κύριο Καρδόνα. Αυτό που θα κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε σύμφωνα με τους στόχους που έχει καθορίσει η μελέτη θα αρχίσουμε με μια εξήγηση σχετικά με το πρόβλημα της διαφθοράς στις δημόσιες προμήθειες. Τη διαφθορά, όπως είπα. Μετά θα συζητήσουμε ορισμένες καλές πρακτικές γενικότερα και μετά κάποια καλά παραδείγματα που έχουν ακολουθήσει οι χώρες μέλη. Και μετά από αυτό ο Φρανσίσκο Καρντόνα θα παρουσιάσει κάποιες προκαταρκτικές συστάσεις πολιτικής και μετά θα μπορέσετε εσείς να θέσετε ερωτήσεις. Η μεθοδολογία της μελέτης βασίστηκε σε μια έρευνα που κάναμε μεταξύ αξιωματούχων αρμοδίων για δημόσιες προμήθειες για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Εξετάσαμε και την βιβλιογραφία καθώς και προτάσεις άλλων διεθνών οργανισμών και οργανώσεων για να χρησιμοποιήσουμε μια evidence-based approach Μπορούμε λοιπόν να σας δώσουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Πρώτον, για την κατανόηση του φαινομένου της διαφθοράς της δημόσιας προμήθειας πρέπει να πει κανείς ότι είναι δύσκολο να οριστεί αυτή η διαφθορά. Υπάρχουν παρατυπίες, υπάρχουν και δραστηριότητες που είναι πραγματικά εγκληματικές. Υπάρχει και διαφορά της ποινικοποίηση στις χώρες μέλη, καθώς και υπάρχουν και διαφορετικές μορφές διαφθοράς στις χώρες μέλη. Μία από τις βασικότερες μορφές διαφθοράς που είδαμε όπως η δωροδοκία, μετά υπάρχουν πρακτικές απάτης, δηλαδή ε, απατηλή εμφάνιση ή παρουσίαση ορισμένων ε, γεγονότων σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Είδαμε συμπεγνία μεταξύ προσφερόντων και δημόσιων αξιωματούχων για να κινήσουν τη διαδικασία προς μια κατεύθυνση ενός δηλαδή παίκτη, ενός operator. Είδαμε επίσης δραστηριότητες όπου οι προσφέροντες παρακολύουν άλλους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν προέρχονται από διάφορες οργανώσεις, από μη κρατικές οργανώσεις, από την Transparency International, επίσης από εθνικές αρχές που έχουν εντοπίσει παρατυπίες όπως ε, φορολογικές αρχές, τα ελεγκτικά συνέδρια, ο ΟΣΑ επίσης σε διάφορες φάσεις των διαδικασιών. Όταν για παράδειγμα γίνεται η αξιολόγηση των αναγκών που είναι η αρχική φάση της δημόσιας προμήθειας όπου λαμβάνεται η απόφαση σχετικά με το αντικείμενο της ε, προμήθειας, καθώς επίσης καθορισμός και του προϋπολογισμού. Είδαμε ότι αυτός ο τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος, γιατί συμβαίνει καμιά φορά οι συμβάσεις να δίνονται στη βάση συμφερόντων πρώην αξιωματούχων που ευνοούν επίσης κάποια πολιτική τοποθέτηση. Μετά προχωρούμε στη φάση όπου αρχίζει, είναι η φάση πρώτων προσφορών, όπου δηλαδή οι αρχές εκκινούν την διαδικασία. Και εκεί η διαφθορά λαμβάνει διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι δωροδοκούνται για να γράψουν με τέτοιο τρόπο την ε, ε, πρόσκληση εκδήλωση προσφορά που να ταιριάζει στα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου προσφέροντος. Υπάρχουν και άλλε δυνατότητες. Γίνεται κατάχρηση της άμεσης ανάθεσης, για παράδειγμα. Για να μπορεί να γίνει άμεση ανάθεση σε κάποιον operator, εφόσον δεν φτάνει σε ένα κατόφλι, τότε κατατέμνουν την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος σε κομμάτια, ώστε να μην ξεπερνάει το κατόφλι που προβλέπει ο νόμος. Επίσης, πολλούν την επιρροή τους, δηλαδή ορισμένοι μπίντερ, ορισμένοι προσφέροντες λαμβάνουν το κείμενο της ε, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πριν από τους άλλους. Επίσης, στην ανάθεση των συμβάσεων βλέπουμε διάφορες μορφές διαφθοράς. βλέπουμε επηρεασμό των ε, όσων ε, λαμβάνουν τις αποφάσεις, σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης η αξιολόγηση των προσφορών δεν γίνεται δημοσία, ώστε όσων οι προσφορές απορρίπτονται είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουν γιατί και να μπορέσουν να αντιδράσουν. Στην φάση εφαρμογής της σύμβασης που μπαίνει δηλαδή η η διαδικασία όταν υπογραφεί η προσφορά, ε, όταν υπογραφεί η ανάθεση μάλλον, συχνά είναι πολύ χαμηλής ποιότητας η, ε, το αγαθό ή η υπηρεσία που προσφέρει ο προσόν έγινε ανάθεση. Συχνά οδηγούνται σε εκ νέου διαπραγμάτευση, ώστε επέρχονται τότε σημαντικές αλλαγές στην αρχική σύμβαση. κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστου. Το νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης σε αυτό πρέπει να τονιστούν δύο πράγματα. Αφενός το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες αναθέσεις, δημόσιες προμήθειες στοχεύει κυρίως στη διευκόλυνση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Αυτό είναι πραγματικά μοναδικό φαινόμενο, διότι συνήθως αυτά εναπόκεινται στη διακριτική ευχαίρεια των χωρών μελών. Είναι κοινοτικό κεκτημένο πρέπει να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες και έχει σημαντική επιρροή στις δημόσιες διοικήσεις των χωρών μελών. Οι βασικές οδηγίες είναι η κλασική Utility Directive, η οι οποίες οδηγίε αυτές θεσπίζουν κριτήρια που οφείλουν οι χώρες μέλη να εφαρμόζουν στις πολιτικές δημοσίων προμηθειών στο εθνικό επίπεδο. Εμείς έχουμε κάνει και ένα ιδιαίτερο σημείωμα για τις προμήθειες άμυνας, όπου είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε διαφθορά. Διότι εκεί δαπανούν οι χώρες πολλά χρήματα Επίσης η οδηγία περί μέσων, ενδίκων μέσων δηλαδή, είναι πολύ σημαντική, Remedies Directive, για να ρυθμίζει τη διαδικασία και είχε σημαντική επίπτωση στο εθνικό επίπεδο. Είδαμε, εξετάζοντας τις διαφορές χώρες μέλη, ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας έχει ολοκληρωθεί σε μέγα βαθμό. Υπάρχουν ορισμένε παραβιάσεις. Υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις ορισμένες φορές στα εθνικά δίκαια. Για παράδειγμα, για το μηχανισμό επανεξέτασης, όταν δηλαδή γίνεται προσφυγή κατά τμήματος της διαδικασίας, τότε υπάρχουν και ένδικα αλλά και άλλα μέσα προσφυγής. Οι διεθνείς κανόνες για τις δημόσιες προσφορές, για τις δημόσιες αναθέσεις και προμήθειες έχουν ενδιαφέρον λόγω του γεγονότος ότι στηρίζουν την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, τη λειτουργία της δηλαδή, επιτρέπει όμως και σε οικονομικούς operator από την Ευρώπη να έχουν πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών. Οι, σημαντικότεροι διεθνείς κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, άλλες διεθνείς συμβάσεις του ΟΣΑ για παράδειγμα, σημαντικό εργαλείο το οποίο έχει ποινικοποιήσει την δωροδοκία αλλοδαπών αξιωματούχων. Επίσης, ορισμένα σημαντικές, ορισμένες σημαντικές διατάξεις περί έξω εδαφικότητας, ετεροδικίας δηλαδή, περί ετεροδικίας, που εκεί επιτρέπουν να λαμβάνονται μέτρα κατά διαφορά και μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτή η ετεροδικία σημαίνει ότι οι εταιρείε οφείλουν, αφού είναι αμερικανική νομοθεσία αυτή, να σέβονται τον νόμο έστω και αν δραστηριοποιούνται αλλού, αλλά εφόσον έχουν κάποια διασύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και το Government Procurement Act, νόμος περί κρατικών προμηθειών, που θεσπίζει ορισμένα πρότυπα, για παράδειγμα τη δημιουργία ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού. Υπάρχει και ένα άρθρο στη Γενική Συμφωνία περί για να γίνει η συζήτηση στις δημόσιες προμήθειες διεθνώς. Ε, συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται στοχεύουν κυρίως αναφέρονται στην πλήρωση αυτού, αυτής της αρχής, στην εφαρμογή αυτής της αρχής στις διεθνείς δημόσιες προμήθειες. Τώρα, αντιμετωπίσαμε και ορισμένες προκλήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά την μέτρηση του κόστους της διαφθοράς. Η δυσκολία βέβαια εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πληροφορίες που να επιτρέψουν συγκριτικές μελέτες για την διαφθορά. Είδαμε ότι οι πιο αξιόπιστες μελέτες είναι ορισμένες οι οποίες αναλύουν ολόκληρα συστήματα, εντοπίζουν τις αδυναμίες και εντοπίζουν κινδύνους διαφθοράς. Γιατί με τη διαφθοράς θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, άμεση αξιολόγηση συγκεκριμένων έργων. Οι αδυναμίες του συστήματος, η πρώτη ε, φάση, pre-bidding δηλαδή και η post-bidding, Εκεί οι κύριες αδυναμίες, όπως εντοπίσαμε στην έκθεσή μας, εντοπίζονται στην φάση πρώτων προσφορών, όπου υπάρχει πολλή διάδραση μεταξύ πολιτικών και συμβούλων, διαφόρων εταιριών συμβούλων, που καλούνται να αξιολογήσουν τις ανάγκες της δημόσιας προμήθειας. Άρα πρέπει να είναι επαρκής η αξιολόγηση των ε, αναγκών, καθώς επίσης πρέπει να είναι επαρκής η αξιολόγηση των βάσεων για τον προϋπολογισμό. Μετά μπορεί να υπάρχει στην επόμενη φάση, ε, μπορεί να υπάρχουν αδυναμίες στην έγκριση, στη ε, διαδικασία έγκρισης, άλλες προκλήσεις στις δημόσιες προμήθειες, βασικές προκλήσεις δηλαδή, που αντιμετωπίσαμε μέσα σε ιδιωτικές εταιρείες, είναι πολιτικά πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό και καμιά φορά χρησιμοποιούμε τέτοια, τέτοιες σχηματικές παραστάσεις για παράδειγμα για παροχή ε, ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού όπου υπάρχει δηλαδή οικονομικό συμφέρον του ιδιωτικού τομέα και βεβαίω και ανάληψη κάποιου επιχειρηματικού κινδύνου αφού προβαίνουν σε επενδύσεις οι εταιρείε αυτές. Κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι αν υπάρχουν σκάνδαλα υφίσταται μεγάλη ζημιά η αξιοπιστία. Η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού θα έχει επίδραση στην απασχόληση. Ταυτόχρονα ένας υπερεθνικός οργανισμός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τον στόχο, έχει τον σκοπό να διευκολύνει και να ανοίξει και διεθνείς αγορές δημοσίων προμηθειών για χάρη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Υπάρχουν και προκλήσεις στην ε, συνεργασία μεταξύ αξιωματούχων αρμοδίων για τις ε, προμήθειες και είναι και ένα ζήτημα λογοδοσίας εκεί γιατί μεταφέρονται από εκλεγμένους, από ερετούς ε, πολιτικούς άρχοντες αρμοδιότητες στους αξιωματούχους που είναι αρμόδιοι για τις διαδικασίες. Α, δεν μου μένει χρόνος. Καλά το καλύτερο τότε είναι να δώσω τον λόγο στον Φρανσίσκο Καρδόνα. Ευχαριστώ. Εγώ μόνο για να, να πω λίγα λόγια για να ολοκληρώσω και να σας μιλήσω για τις ε, προσωρινές ε, συστάσεις οι οποίες μας απασχολούν ακόμα και νομίζουμε ότι θα χωρίσουμε τις συστάσεις σε δύο βασικούς τομείς. Καταρχήν την καταστολή της διαφθοράς της δημόσιας προμήθειας και της, ε, την πρόληψη. Ως προς την πρόληψη ε, ακολουθούμε την λογική της οδηγίας περί δημόσιων προμηθειών για να δημιουργήσουμε μία εννέα αγορά και γι' αυτό χρειάζεται ένας και μοναδικός νόμος ε, για τις ε, δημόσιες προμήθειες, όπως είπε και ο συνάδελφος, αλλά ακόμα δεν έχουμε το ίδιο ποινικό, δεν μας διέπει το ίδιο ε, ποινικό σε σχέση με τη διαφθορά και τα διάφορα αδικήματα. Γι' αυτό και δημιουργείται η αρχή του Ευρωπαίου Ισαγγελέα που προβλέπεται για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας τομέας λοιπόν όπου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ως προς την πρόληψη θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη και τις βέλτιστες πρακτικές και θα μπορούσαμε να προτείνουμε και προσωρινές λύσεις. Χρειαζόμαστε καλύτερους κανόνες, για ιδιαίτερα ως προς την σύγκρουση συμφερόντων, διακρίνοντας μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και πολιτικών διότι τα συμφέροντα δεν είναι ίδια μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών όταν μιλάμε για δημόσιες προμήθειες. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει ένα σκοτεινό τομέας που αφορά τη διαδικασία πριν από το διαγωνισμό, δηλαδή την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Είναι ένας τομέας ο οποίος ε, δεν διέπεται από κανόνες, γίνεται πολιτική συζήτηση, κάτι το οποίο είναι θετικό, αλλά υπάρχει διακριτική ευχέρεια η οποία απορρέει από περίεργους κανόνες και συμφέροντα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα no man's land εδώ. Είναι στο που δεν διέπεται από κανόνες και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε την διαφθορά και ένα γενικό συμπέρασμα που αφορά ολόκληρο, τομέα, ολόκληρο το τομέα των δημόσιων προμηθειών είναι η διαφάνεια. Είναι μία αρχή, μία βασική αρχή που θα πρέπει να διέπει όλους τους κανονισμούς. Όσο περισσότερη διαφάνεια υπάρχει, τόσο λιγότερη είναι η διαφθορά. Αυτές είναι οι κεντρικές ιδέες που διέπουν την εργασία μας. Βλέπουμε την εμπειρία των κρατών μελών και τα δεδομένα από τους διεθνούς, διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, το οποίο εργάζεται για την πρόληψη διαφθοράς στον τομέα των προμηθειών της άμυνας. διότι κάθε χώρα ζητά εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα χωρίς να δικαιολογείται άμεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα αρχίσουμε με τον γύρο των ερωτήσεων και τη συζήτηση γενικότερα. Ποιος θέλει το λόγο, Μπορσελίνο. Η κυρία Μπορσελίνο, καλημέρα σας. Θα ήθελα να εκφράσω μία σκέψη. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτά τα περάσματα που κάνουμε, τόσο πιο δύσκολη είναι η διαφάνεια. Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που διαθέτουμε σε αυτό τον τομέα. Πόσο μπορούμε να περάσουμε ε, αυτό το πρόσκομα στις δημόσιες προμήθειες ποια, ποιο είναι και το κατόφλι. Υπάρχει κατόφλι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει στην, ε, ως προς την ευαλωτότητα. Έγινε λόγος και για πρόληψη. Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης ε, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Νιωτοντάν. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και λυπάμαι που περιορίζεστε από το χρόνο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η φύση της δουλειάς μας. Θα μπορούσατε να μας δώσετε παραδείγματα. Λέτε ότι δεν έχουμε τυποποίηση του εγκλήματος όσον αφορά τα εγκλήματα στις διάφορες χώρες μέλη. Ας πούμε, μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα σε ποια χώρα ένα έγκλημα έγκλημα. Δεν θα ήταν έγκλημα σε εκείνη τη χώρα, ενώ σε κάποια άλλη θα θεωρεί το πολύ σοβαρό έγκλημα. Δεύτερον, έχω την υποψία ότι ακόμα και αν καταλήξουμε στο ότι κάποιο σε μια χώρα μέλος έχει καταχραστεί κοινοτικών κονδυλίων, πώς θα διωχθούν σε εθνικό επίπεδο. Γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές φυλακές. Πώς γίνονται λοιπόν αυτές οι διώξεις, γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σπάνιες, πώς. Η κυρία Τάνια Φαγιών. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα, οπότε ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη αν σας ρωτήσω κάτι το οποίο έχει ήδη απαντηθεί. Θέλω να σας ζητήσω λεπτομέρειες για τις συστάσεις σας, πώς η πολιτική θα λογοδοτούν περισσότερο, θα είναι περισσότερο υπεύθυνοι, θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Υπάρχει μια προσωρινή έκθεση της Επιτροπής ΚΡΙΜ που το αναφέρει και γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια περιπτώσεις διαφθοράς στο δημόσιο τομέα που έχει τεράστιες επιπτώσεις ως φαινόμενο σε όλο το δημόσιο τομέα και βέβαια στους υπεύθυνους πολιτικούς. Τουλάχιστον πέντε χρόνια ε, θέλουμε ποινή για όσους... Μάλλον χρειάζονται πέντε χρόνια για να καταλήξουμε ε, σε περίπτωση που έχουμε ύποπτους πολιτικούς για διαφθορά. Έπειτα υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Πώς πιστεύετε εσείς ότι μπορούμε καλύτερα να καταστήσουμε υπεύθυνου τους πολιτικούς. Γνωρίζουμε περιπτώσεις πρόσφατα στη Σλοβενία, όπου το δικαστήριο καταλήγει για πολιτικούς υψηλά ιστάμενους, ενώ μετά δεν δίνεται καμία συνέχεια. Πώς λοιπόν θα έχουμε ένα δικαστικό σύστημα επίσης με μεγαλύτερη διαφάνεια, ανεξαρτησία. Πιστεύετε δηλαδή ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση ή υπάρχει περιθώριο για παρετέρω Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρόνα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καταλάβω αυτή την πτυχή του θέματος γιατί μιλήσατε για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Με βάση τη δική σας εμπειρία θα ήθελα να σας ρωτήσω Ποια είναι τα κράτη τα οποία είναι πιο υπεύθυνα στον τομέα της διαφάνειας ε, ως προς τους ε, δημόσιους διαγωνισμούς και ποια κράτη δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Ζόντεργαρντ. Σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση όσον αφορά τα όρια των προσφορών για προμήθειες. Και είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό, διότι υπάρχουν πολλά σημεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί δήμοι, που χρησιμοποιούν πολύ σημαντικά κονδύλια για να ανταποκριθούν σε προσφορές που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς τελικά να ενδιαφέρεται κανείς πρέπει πιστεύετε να πάμε σε αύξηση του ορίου των προσφορών για προμήθειες χωρίς να υπάρξει κατάχρηση οργανωμένο έγκλημα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Έπειτα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το φαινόμενο της υπεργολαβίας. Ας πούμε ότι έχουμε μία επιχείρηση που παίρνει ένα συμβόλαιο και το οποίο μετά το κόβουμε σε κομματάκια και το δίνουμε σε άλλες μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο φαινόμενο πρέπει να απαγορευτεί? Να πούμε ότι όσοι, αυτοί μάλλον που κάνουν την καλύτερη προσφορά, αυτοί πρέπει να εκτελέσουν και το έργο. Δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Και έρχομαι και στην τελευταία μου ερώτηση. Σχετικά με το υλικό των προσφορών. Δεν ξέρω αν τον μελετήσατε αυτό στην έρευνά σας, στη μελέτη σας. Αλλά εδώ λοχεύει ένας κίνδυνος σε σχέση με το υλικό αυτό. Θα μπορούσε να τύχει κατάχρησης. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μια δομή του υλικού αυτού η οποία να είναι πιο προστατευμένη, πιο διαρθρωμένη έτσι ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για καταχρήσεις. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής μας, οι εισηγητές μας μάλλον, πρώτα απ' όλα ο κύριος Μπέκ και μετά ο κύριος Καρδόνα. Ο κύριος Μπέκ λοιπόν πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές που θίξατε και εσείς. Μία από τις πτυχές που αναφέρθηκε είναι το γεγονός ότι ένας πιο μεγάλος χώρος είναι πιο ευάλωτος. Οι... Τα διάφορα στάδια όμως ελέγχονται από ρυθμιστικές αρχές. Το στάδιο της προσφοράς για παράδειγμα έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις για τις προμήθειες. Μόλις υπάρξει η υπογραφή, τότε αμέσω αρχίζει και ισχύει ο νόμος για τις συμβάσεις. Βέβαια, στο προηγούμενο στάδιο, πριν την προσφορά, δεν έχουμε πολλά περιθώρια να δράσουμε και να αποφύγουμε τη διαφθορά. Το κύριο θέμα είναι η γραφειοκρατία, ο περιορισμό τη γραφειοκρατίας στι κρατικέ προμήθειε είναι πολύ βασικό. Είναι κάτι θεμελιώδε για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερα περιθώρια για διαφθορά. Οι μελέτη μα και άλλε μελέτε που έχουν παρουσιαστεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην υπερβολική γραφειοκρατία και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, από την και τον έλεγχο από την άλλη. Άρα όσο πιο πολύ γραφειοκρατία έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι για κάποιον να προχωρήσει σε διαφθορά. Η γνώμη μου για αυτό το θέμα είναι ότι χρειάζεται θεσμική ενίσχυση σε επίπεδο χωρών μελών, να γίνει ανάλυση και το θεσμικό πλαίσιο να ενισχυθεί, να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να γίνουν συστάσεις για την ενίσχυση του θεσμικού αυτού πλαισίου. Είναι καλό δηλαδή να γίνει μια αξιολόγηση στις χώρες μέλη. Στο θέμα της διαφθοράς λέμε ότι ο κόσμος προχωράει σε διαφθορά εφόσον το σύστημα του επιτρέπει τη διαφθορά. Όσον αφορά τα όρια τώρα. Είναι κάτι περίπλοκο γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο όριο που βασίζεται σε εκτιμήσεις του ενός πέμπτου των προμηθειών που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις προμήθειες. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα του ορίου, πρέπει να βασιστούμε στην ακαιρεότητα των αρχών στα κράτη-μέλη που είναι αρμόδιες για τις προμήθειες. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να διευκολύνουμε ένα δίκτυο γνώσης για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης μεταξύ των χωρών μελών για να γνωρίζουν πώς καλύτερα μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις. Ρωτήσατε για τη δίωξη της διαφθοράς. Είναι περίπλοκο ζήτημα αυτό και είναι περίπλοκο γιατί όπως είπαμε και πριν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφές διαφθοράς στις διάφορες χώρες. Κακή επιρροή. Στη Γαλλία είναι κάτι που δεν διώκεται ως έγκλημα. Για παράδειγμα. πρέπει να ενισχυθεί δίωξη στις χώρες μέλη, καταρχήν. Και έχουν υπάρξει στην Ισπανία, για παράδειγμα, πρωτοβουλία για την ε, δίωξη σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Ο εισαγγελέα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητος. Ορισμένοι προτιμούν να είναι αυτός ο οποίος ηγείται τον ανακρίσιο της αστυνομίας. Άλλοι δεν το θέλουν αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πόσες τέτοιες περιπτώσεις διώξεων διαφθοράς έχουμε, είτε γιατί δεν ανακοινώνονται, είτε γιατί είναι δύσκολη η σύγκριση. Και το θέμα είναι, οδηγεί σε κυρώσεις η δίωξη αυτή. Υπάρχει πολλές φορές ατιμορρησία της διαφθοράς. Κάτι το οποίο βέβαια έχει τεράστιες επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Γιατί όταν οι πολίτες βλέπουν ότι στο τέλος ε, μία διαφορά δεν τιμωρείται, έχουν την τάση να ζητούν επίκαια. Το κοινό λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφθορά στο δημόσιο τομέα δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά. Ένα άλλο θέμα είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αλλά εδώ ο συνάδελφος θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, ναι, θέλω και εγώ να θίξω κάποια ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Το θέμα της εναρμόνισης πρώτα απ' όλα. Η εναρμόνιση δηλαδή της νομικής περιγραφής του εγκλήματος στον ποινικό κώδικα. Είναι αλήθεια ότι διαφέρει από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που κάνει πιο δύσκολη την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Την δίωξη της εγκληματικότητας, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η διαφορά στην νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τις προμήθειες. Ρωτήσατε κύριε Κορώνα, ποιες χώρες θα μπορούσαμε να προτείνουμε ως παράδειγμα, όχι επειδή είσαστε Ιταλός, αλλά νομίζω ότι η Ιταλία έχει κάνει τεράστια βήματα σε αυτό. Διότι έχουν ένα πολύ περίπλοκο πρόγραμμα όσον αφορά τις διαδικασίες καταπολέμησης της διαφθοράς πώς αντιμετωπίζετε το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει επίσης ένα πολύ καλό σύστημα κατάσχεσης των προϊόντων διαφθοράς. Αυτό είναι ένας από τους μηχανισμούς ο οποίος τελικά πλήττει περισσότερο αυτούς που δραστηριοποιούνται στη διαφθορά. Η κατάσχεση δηλαδή. Θέλω να κάνω και κάποιο σχόλιο για αυτό που είπε η κυρία Φαγιόν για το πώς μπορούμε να απαιτήσουμε από τους πολιτικούς να λογοδοτούν περισσότερο και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ξέρετε, οι κρατικές προμήθειες χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες ως κύρια πηγή χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτό πρέπει να το πούμε. Τώρα, πώς το αντιμετωπίζει κανείς αυτό το ζήτημα. Το θέμα αυτό το έχουμε αφήσει εκτός της μελέτης μας γιατί είναι περίπλοκο και χρειαζόταν πολύ περισσότερη προσπάθεια και χρόνο που δεν διαθέταμε. Πέρα όμως από τους περιορισμούς, από την εφαρμογή όλων των μηχανισμών, των ελέγχων κτλ, ίσως θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την διάκριση Τη πολιτική δραστηριότητα από τη διοικητική δραστηριότητα. Γιατί μερικέ φορές έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε διοικητικού μηχανισμούς για να ελέγξουμε τους πολιτικούς. Ενώ συγχρόνω οι πολιτικές αποφάσεις βρίσκονται εκτός διοίκηση. και η διοίκηση εφαρμόζει τις πολιτικές αποφάσεις. Είναι δηλαδή δύο κόσμοι που θα έπρεπε να χωριστούν. Ίσως να είναι ένα πεδίο μελέτης από το οποίο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Όμως προς το παρόν, παρόλο που θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, δεν έχουμε τους μηχανισμούς να το λύσουμε. Έχουμε παραδείγματα από διάφορα κοινοβούλια, έχουμε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, από τη Βουλή, όπου υπήρξαν κάποια φαινόμενα διαφθοράς, δυσάρεστα. Έχουμε κάποια εμπειρία, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιο συστημική, συστηματική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε γενικά συμπεράσματα, άρα να προτείνουμε και συγκεκριμένες λύσεις. Ένα σχόλιο ακόμα επιτρέψτε μου για την υπεργολαβία, που είπαμε ότι είναι μία από τις αδυναμίες της διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε ότι από τη στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της διαδικασίας που προβλέπεται από την οδηγία για τις συμβάσεις. Γιατί είναι τότε που αποφασίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ελέγχουμε και από εκεί και πέρα η διαδικασία εμπίπτει στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή που υπάρχει η σύμβαση, όμως η εφαρμογή της βρίσκεται εκτός πεδίου εφαρμογής της οδηγίας αν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιήσουν υπεργολαβία και τελικά η ποιότητα που προσφέρουν δεν είναι αρκετή, αρκετά ικανοποιητική, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ενώ αν προβλέπετε κάτι σχετικό στους όρους της σύμβασης, τότε ναι, μπορούμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο μιλητές Μπέκε και Καρδόνα για αυτές τις άκρος ενδιαφέρουσες πληροφορίες αν και είναι γεγονός ότι τα θέματα αυτά αφορούν την ΚΡΙΜ αλλά και τον ρόλο της πολιτικής. Θεωρώ ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη αποφασιστικότητα γιατί ότι βλέπουμε ότι στη δημόσια διοίκηση υπάρχει διαφθορά, κάτι το οποίο είναι ολέθριο, για την εικόνα των κοινοτικών οργάνων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την διαθέσιμότητά σας και τώρα περνάμε στο δεύτερο κλάστερ που είναι οι διεθνείς έρευνες και οι συνέπειες αυτών σε σχέση με τις εγκληματικές ενέργειες του Ντάουσμπουργκ στη Γερμανία. Θα ακούσουμε τον Ραλφ Ράινερ Γέγκερ, ο οποίος θα μας μιλήσει και άλλους δύο ομιλητές, τον Νικόλα Γκρατέρη που θα μας μιλήσει για την διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση της φαγής του Ντάουσμπουργκ και τέλος ο Γιούργεν Ρότ, ο οποίος είναι ένας ερευνητής στη Φραγκφούρτη και θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις της Ιταλικής μαφίας στη Γερμανία και τις επιπτώσεις της φαγής στο Ντάουσμπουργκ. Ο κάθε ομιλητής έχει 12 με 13 λεπτά στη διάθεσή του και δίνω το λόγο στον Ρολφ Ράινερ Γέγκερ καταρχήν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τη νύχτα της 15ης Αυγούστου 2007 οι φόνοι που έγιναν στο Ντουισμπουργκ τάραξαν τα νερά στη Γερμανία. Σκοτώθηκαν, σκότωσαν έξι νεαρούς μετά από μια γιορτή γενεθλίων σε ένα ιταλικό εστιατόριο μέσα στο κέντρο του Ντουίσπουρ. Πραγματική εκτέλεση από δύο πυροβόλα όπλα. Και φαίνεται πως υπεύθυνη ήταν η καλαβρέζικη οργάνωση της μαφίας Ντρανγκέτα. Ο, Ιταλικό, ο Ιταλός Υπουργός των Εσωτερικών μίλησε αμέσως μετά για βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών στο Σαν Λούκα. Οι γερμανικές αρχές και η δική μας αστυνομική διεύθυνση Duisburg γνώριζαν περί της βεντέτας αυτής. Ωστόσο δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με το ότι η βεντέτα αυτή θα μπορούσε να μεταφερθεί στη Γερμανία ή ακόμα πιο συγκεκριμένα στο Duisburg οι γερμανικές αστυνομικές αρχές εντυπωσιάστηκαν από την αγριότητα του εγκλήματος και την αδιαφορία απέναντι στο υψηλό αριθμό των θυμάτων, αδιαφορία πλευράς των δραστών. Φοβηθήκαμε μιμητισμό, αντεκδικήσεις και άλλες τέτοιες πράξεις επίλυσης συγκρούσεων των μαφιών στην ε, ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία, που μέχρι, μέχρι τότε δεν είχε πολλά τέτοια φαινόμενα. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καταπολέμησης του Εγκλήματος στην διαρρεύνηση υποθέσεων της Ιταλικής Μαφίας και των διαφόρων υποδιαρέσεών της φάνηκε καθαρά ότι είχε υποστεί μείωση προσωπικού. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε πολλά κρατήδια της Γερμανίας δεν είχε στραφεί τόσο πολύ σε ομάδες της μαφίας. Η ε, γερμανική αστυνομία θεωρούσε μεν ότι η μαφία χρησιμοποιεί την γερμανική ε, επικράτεια ως χώρο καταφυγής και επενδύσεως ε, ε, κεφαλαίων από εγκληματικέ δραστηριότητες δεν είχαν σημειωθεί όμως σημαντικές επιθέσεις, εκβιασμοί, απαγωγές κλπ. Φάνηκε όμως καθαρά με το παράδειγμα αυτό του Ντουίσπουργκ ότι η μαφία δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Οι Ιταλοί εισαγγελείς που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων της μαφίας είχαν προειδοποιήσει απέναντι στο ενδεχόμενο τέτοιων δραστηριοτήτων και στη Γερμανία. Οι δικές μας έρευνες έδειξαν ότι οι γνώσεις μας για τις ομάδες μαφίας και για την δράση τους ήταν απλά στοιχειώδεις. Δεν είχαμε καμία συστηματική συλλογή στοιχείων για την ε, μαφία. Έτσι εκλήθη η πολιτική να δράσει. Ο πρόεδρος του ΜΠΚΑ, της υπηρεσίας μας δηλαδή, μετέβη στην Ιταλία, υπέγραψε συμφωνία για τη δημιουργία μιας task force για την συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τις εγκληματικές δραστηριότητες των Ιταλών μαφιόζων στην Γερμανία. Ταυτόχρονα οι γερμανικές αρχές θα διεβίβαζαν τις δικές τους πληροφορίες από τις έρευνές τους στους Ιταλούς αξιωματούχους. Οι Ιταλοί είχαν και φαίνεται πως έχουν ακόμη την ανησυχία ότι και στην ε, ε, γερμανική αστυνομία υπάρχουν μη στεγανές, ε, υπάρχουν κάποια μη στεγανά και διστάζουν να δώσουν πληροφορίες στους Γερμανούς για να μην θέσουν σε κίνδυνο τις δικές τους έρευνες. Ωστόσο αποκαταστάθηκαν κάποιες προσωπικές επαφές και παρόλα αυτά φάνηκε ότι οι εγκληματολόγοι των δύο χωρών ε, καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε πολύ διαφορετικά δικαιικά συστήματα. Η καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας της ε, μαφίας στην Ιταλία είναι μοιρασμένη σε υπηρεσίες όπως Πολιτσία Διστάτο, Καραμπινιέρι, Guardia di Finanza και άλλες υποδιαρέσεις των αρχών αυτών. Μόνο η Γενική Εισαγγελία έχει συνολική επισκόπηση όλων των διαδικασιών αυτών και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών αυτών είναι μάλλον η εξαίρεση. Και η ανάγκη τήρησης μυστικότητας απορρίτου φαίνεται πως υπερέχει. Και πιθανότατα υπάρχουν και λόγοι. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί εγκληματολόγοι έμαθαν ότι δεν ενδιαφέρονται οι Ιταλικές διοκτικές αρχές τόσο πολύ για την διευκρίνηση ενός έστω και εξαπλού φόνου, αλλά τους ενδιαφέρουν περισσότερο οι συνολικές εγκληματικές δραστηριότητες μιας ομάδας που κρατούν και πολλά χρόνια με την παρακολούθηση τηλεφώνων, επικοινωνιών και εντός και εκτός κατοικιών σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο χ, στη βάση των, των μη αποδείξεων, προχωρούν τότε σε αριθμό ε, συλλήψεων και κατασχέσεων. Οι έρευνες λοιπόν που διεξάγονται από τις Ιταλικές Αρχές έχουν περισσότερο στόχο να καταστήλουν την εγκληματική δραστηριότητα μιας οργάνωσης για, μακρότερο χρονικό, ε, για μακρότερη χρονική περίοδο. Έτσι, καμιά φορά δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην ανάγκη ε, συνεργασίας με άλλες ε, διοκτικές αρχές στην ε, Ευρώπη. Εν ώψη λοιπόν του γεγονότος αυτού, η task force για την οποία μίλησα δεν ανταποκρίθηκε στις ε, προσδοκίες μας. Οι γερμανικές ε, ανακριτικές αρχές δεν έλαβαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την Ιταλία. Ενώ η Ευρώπη, και αυτή είναι η σύστασή μας προς εσάς, έχει κάθε συμφέρον να δραστηριοποιηθεί για μια πανευρωπαϊκή συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, όχι μόνο για την Ιταλική μαφία, αλλά για παράδειγμα για ε, διαρρήκτες Κόσοβο-Αλβανούς, για Λιθουανούς ε, κλέφτες, για άλλους διαρρήκτες από Ρουμανία, Βουλγαρία, για απάτες, για ε, απάτες από ε, ομάδες απαταιώνων μάλλον από διάφορες χώρες όπως και Πολωνία, Ρουμανία κλπ. Και αυτά να γίνουν σε μια σε ένα επίπεδο διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών. Ένα θετικό πράγμα που προέκυψε είναι ότι η Ιταλία απέστειλε οι δήμονες από το Σαν Λούκα στη δική μας αντιεκκληματική υπηρεσία για να μπορέσουν να αρχίσουν έρευνες και στην Ιταλία. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν, όπως θέλαμε στην αρχή, να φτιάξουμε μια κοινή ερευνητική ομάδα που σύμφωνα με την σύμβαση του ΠΡΙΜ που είναι διεθνής σύμβαση 11 ευρωπαϊκών ε, χωρών μελών και της Νορβηγίας θα επέτρεπε τη συνεργασία αυτή. Από ό,τι ξέρω δεν εφαρμόζεται ακόμα η σύμβαση του ΠΡΙΜ στην Ιταλία, κάτι το οποίο προκαλεί προβλήματα στη συνεργασία, ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα. Η συνεργασία στα Joint Investigation Team που συνοδεύεται και από την Ευρωπόλ από την αστυνομική πλευρά και την Eurojust από την ε, πλευρά των δικαστηρίων είναι ο δρόμος που υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Από την άποψη της δικής μας ε, επαγγελματικής οργάνωσης θεωρούμε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε τις πληροφορίες που έρχονται από τα διάφορα δικαιϊκά συστήματα και οι ανακρίσεις να μην γίνονται πλέον μόνο εγχώρια, αλλά πανευρωπαϊκά. Η σύμβαση του πριν προβλέπει ότι οι αστυνομικές και άλλες διοκτικές αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα και τραπεζικά των ε, συμβαλωμένων χωρών, καθώς επίσης και σε τράπεζες δεδομένων DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων, και σε άλλα έγγραφα, επίσης αυτοκινήτων κλπ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτή η πολύ σημαντική σύμβαση του ΠΡΙΜ δημιουργεί και τις τράπεζες δεδομένων DNA με το προφίλ DNA των δραστών γιατί υπάρχουν και δράστες οι οποίοι είναι άγνωστοι στις αστυνομικές αρχές επιτρέπει λοιπόν την διεθνή ενεργασία και οργάνωση εδώ εξ όσων γνωρίζουμε στην Ιταλία υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις δεν υπάρχει καν ακόμη μια κεντρική τράπεζα δεδομένων για το DNA των εγκληματιών. Και στην Ομοσπονδιακή Γερμανία υπάρχει άνω του ενός εκατομμύριου, άνω του ενός εκατομμυρίου ε, δεδομένα. Σήμερα η απόδειξη στη βάση του DNA είναι η πιο σημαντική και η πιο επιτυχής δυνατότητα απόδειξης των ε, εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αν είχε η Ιταλία το 2007 την Τράπεζα Δεδομένων, DNA, τότε θα ήταν πολύ ευκολότερη και ταχύτερη η διαλεύκανση του εξαπλού φόνου του Duisburg. Θα πρέπει λοιπόν να επιτραπεί η συλλογή στοιχείων DNA. Φαίνεται όμως στην Ιταλία να είναι ακόμα πολύ πιο εύκολο να επιτραπεί η παρακολούθηση τηλεφώνων, η οικειών κτλ. παρά η συλλογή ε, στοιχείων DNA. Έτσι λοιπόν η αστυνομική διεύθυνση του Ίσπουργκ δεν είχε τα δεδομένα αυτά. Ούτε και τρεις εβδομάδες μετά από την ε, εγκληματική πράξη η αστυνομική αρχή του Ντούισπουργκ διαβίβασε τα στοιχεία ενός υπόπτου και ζήτησε τα δεδομένα DNA του, τα οποία έλαβε 21 μήνες μετά. Ούτε καν τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν είναι συγκρίσιμα, για να μην μιλήσει κανείς καθόλου πλέον για DNA. Επίσης, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων είναι τόσο δυσχερή στην Γερμανία ώστε κανείς από τους εγκληματίες αυτούς δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη τράπεζα δεδομένων πανευρωπαϊκή που να μπορεί να ε, ταυτοποιεί και το DNA και εγκληματιών από χώρες όπως η Ρουμανία, η Ισπανία κλπ. Άλλη δυσκολία που διαπιστώνουμε είναι το γεγονός ότι η Ιταλία δεν έχει τράπεζα δεδομένων ούτε για όπλα, ούτε για πυρομαχικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για κλιματικές πράξεις, κάλικες ε, σφαιρών κλπ. Αυτά ανήκουν σε διάφορες ε, αστυνομικές οργανώσεις στην Ιταλία, οι οποίες δρούν και τηρούν τις τράπεζες αυτές δεδομένων μόνο σε επίπεδο περιφερειών. Γι' αυτό χρειάζονται συλλογικές συγκεντρωτικές τράπεζες δεδομένων για τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει μάλιστα να σκεφτείτε εάν αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ε, δημιουργηθούν, να οργανωθούν ε, συγκεντρωτικά στην Ευρώπη. Στις έρευνες που διεξήχθησαν στο Duisburg διαπιστώθηκε ότι το ε, γερμανικό δικαιικό σύστημα δεν ε, συναρμόζεται με το Ιταλικό, για παράδειγμα, στις ανακρίσεις σε πολλές περιπτώσεις. Η Ιταλική, τα νόμη και η νομολογία, αντιθέτως από τη Γερμανία, απαιτούν πάντοτε να παρίσταται συνήγορος της, ε, της πλευράς που έχει υποστεί τη ζημία. Αυτό δεν υπάρχει στη Γερμανία. Εμείς διαβιβάσαμε έγκαιρα τα δεδομένα. Δεν μπόρεσαν όμως να αξιολογηθούν για το λόγο αυτό. Εδώ χρειάζεται να υπάρξει μια εναρμόνιση των δικαιωτικών συστημάτων, διότι δεν θα είναι δυνατόν να γίνονται τα ανακριτικά αυτά βήματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου ενδεχομένως αργότερα θα διεξαχθεί η ποινική δίκη. Η ευρωπαϊκή πολιτική δικαιοσύνης Οφείλει λοιπόν να εναρμονίσει τις διατάξεις αυτές και στην ποινική διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρχουν και ενιαίες δικονομικές διατάξεις που να επιτρέψουν νέες μορφές της συνεργασίας. και για τρέχουσες ποινικέ έρευνες αλλά και για ε, έρευνες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ομάδες εγκληματολόγων ή αστυνομικών υπαλλήλων που να διαθέτουν και γλωσσικές γνώσεις ώστε να καταστεί δυνατή η διασφάλιση των απορριφτικών στοιχείων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο πανευρωπαϊκά και να, μπορεί, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία σε κάθε ποινική διαδικασία σε οποιαδήποτε χώρα μέλος. Εδώ τονίζω βεβαίως και την ε, πολύ θετική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Καλαβρίας. Οι αποστολές που διεξαγάγαμε στις χώρες που συμμετείχαν στην ε, έρευνα αυτή για πολλούς μήνες βοήθησαν στην αλληλοκατανόηση και αυτό το απέδειξε η υπόθεση αυτή του Duisburg. Τέλος, η εγκληματίες στην Ευρώπη δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να κρατάνε τα πράγματα στα χέρια τους. Δρούν διαμεθοριακά και επομένως πρέπει να βρουν απέναντί τους διαμεθοριακά αρμόδιες αστυνομικέ αρχές οι οποίες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δραστηριότητες αυτές ώστε εν τέλει η διεξαγωγή εγκληματικών πράξεων στην Ευρώπη να καταστεί μη ελκυστική για αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Είμαι ο κύριος ε, Γκρατέρη και εδώ και 26 χρόνια ασχολούμαι με τη δραστηριότητα κατά της Ντράγκετα μέσα στα πλαίσια της Γενικής Εισαγγελίας ε, για την καταπολέμηση της μαφίας. Για να μιλήσω για την σφαγή του Ντάουσπουργκ δεν επρόκειτο ε, μόνο για μία γιορτή, διότι στο πορτοφόλι του ε, ενός σκοτωμένου ε, βρέθηκε μία εικόνα η οποία αποδείκνυε ότι συμμετείχε σε δραστηριότητες της Ντράγκετα. Επίσης, σε αυτή την τοποθεσία υπάρχει η, η εικόνα του, Αγίου, του, του Μιχαήλ του Αρχαγγέλου που είναι η εικόνα της ε, Ντράγκετα, το λογότυπο της ε, Ντράγκετα. Δεν πρόκειται για ένα κοινό ε, μαγαζί, είναι για, πρόκειται για μία τοποθεσία όπου συγκεντρώνονταν τα μέλη της Ντράγκετα. Δέκα χρόνια πριν από τον Ντάουσμπουργκ, το 2007, βρέθηκα στη Γερμανία αρκετές φορές γιατί ερευνούσα τη δραστηριότητα της ε, Ντράγκετα για πάνω από 20 χρόνια και γυρίζω τον κόσμο σε 20 χώρες, Βόρειο Αμερική, Νότιο Αμερική, Αυστραλία και ούτω καθεξής, όπου που ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι προβαίνω σε ανακρίσεις πολλές φορές την εβδομάδα, διότι η Ντράγκετα είναι η πιο ισχυρή μαφία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχει το ιονί μονοπόλιο της ε, κοκαίνης στην Ευρώπη μαζί με τους Ε, Για να γυρίσουμε στο Ντάουσπουργκ. Όταν ε, βρέθηκα στο Ντάουσπουργκ άκουσα τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις όπου οι Καλαβρέζοι μιλούσαν για τις τοποθεσίες αυτές. Και μου ελέγχθη ότι θα πρέπει να ε, παρέμβουμε, διαφορετικά θα υπάρξουν τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν και στην Ιταλία. Η μεγάλη δυσχέρεια για μας για μας τους Ιταλούς, όταν μιλάμε με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές στην Ευρώπη, είναι ότι θα πρέπει να καταστήσουμε κατανοητή την παρουσία της μαφίας, όχι μόνο όταν σκοτώνουν, αν η Ντράγκετα, η Καμόρα και η Κόζα Νόστρα βρίσκονται στην Ευρώπη για ανακυκλώσουν, δείχνει, αυτό καταδεικνύει ότι εκεί που δεν γίνεται μία κλοπή ποδηλάτου γίνεται ανακύκλωση, διότι η πρώτη δραστηριότητα είναι η ανακύκλωση και η πώληση της κοκαίνης. Τελεία και παύλα. Το Ντάουσμπουργκ ήταν ένα ατύχημα και έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό διότι η σφαγή έγινε στις 15 Αυγούστου του 2007. Στις 2 Σεπτεμβρίου η ελίτ της Εντράγκετα επέπληξε τα δύο μέλη της οικογένειας και τους επέβαλε την ειρήνη. Τους είπε δηλαδή δεν σας επιτρέπω πλέον τέτοιες δραστηριότητες στο εξωτερικό διότι μας χαλάτε τις δουλειές. Μετά την σφαγή στο Ντάουσπουργκ η γερμανική και η ολλανδική αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβουν, καθώς και οι γερμανικές δικαστικές αρχές. Ποιες ήταν ε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν. Αρχικά με τη Γερμανία θα πρέπει να πω ότι υπήρξαν δυσκολίες, αλλά εργαστήκαμε πολύ καλά. Πρόκειται για αστυνομικές και δικαστικές αρχές που συνεργάζονται. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, όπως είπε και ο κύριος Γέγκερ, ότι δεν υπάρχει ένα interface, ένα ρυθμιστικό interface. Θα πρέπει δηλαδή να μην χάνουμε χρόνο κάνοντας απλώς σεμινάρια, αλλά να δούμε για αυτή τη διάδραση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εάν η δίκη είχε γίνει όχι στην Καλαβρία αλλά στη Γερμανία θα είχαν αθωωθεί οι υπόδικοι. Εμείς ευχαριστούμε την γερμανική αστυνομία διότι συνεργάστηκε μαζί μας ιδιαίτερα στη, στο αποτύπωμα DNA. Θα ήθελα οι Ιταλοί πολιτικοί και οι Ευρωβουλευτές να επιμείνουν έτσι ώστε η Ιταλία να προσχωρήσει στη συνθήκη του ΠΡΟΥΜ. Δεν είναι δυνατόν διαφορετικό να γίνει κάτι διαφορετικό. Η σύμβαση του ΠΡΟΥΜ είναι πολύ σημαντική. Έχουν μία τράπεζα δεδομένων πολύ ισχυρή. Μπήκαν και η Γερμανία και η Ρουμανία και η Τουρκία. Και έτσι μπορέσαμε να ανοιχνεύσουμε 70 εγκλήματα μόνο με το αποτύπωμα DNA. Είναι πολύ σημαντική η προσχώρηση και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Θα πρέπει να πω ότι δεν ισχύει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τράπεζες δεδομένων στην Ιταλία. Υπάρχουν δύο πλήρως ενημερωμένες ε, των ε, ε, αστυνομικών αρχών, των δικαστικών. Και μπορώ να σας πω ότι η ελίτ των αστυνομικών αρχών της Ιταλίας είναι από τις καλύτερες του κόσμου. Και αυτό το λέω αφού γύρισα όλο τον κόσμο. Όμως στην Ευρώπη, όσο πηγαίνουμε προς βορρά, δεν ε, ανοιχνεύεται η δράση της μαφίας. Και Δυστυχώς η Ευρώπη είναι σαν ένα μεγάλο βοσκοτόπι οποίος μπορεί, όπου οποιοδήποτε μπορεί να δράξει όποια ευκαιρία θέλει. Δηλαδή υπάρχουν μέλη της Ντράγκετα, της Κόζα Νόστρα και της μαφίας που πολλούν κοκαίνη και δεν ελέγχονται. Εγώ βρέθηκα στη Βόρεια Ευρώπη σε ένα κράτος όπου μου είπαν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την τράγκετα γιατί δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Μα αυτό δεν είναι δυνατόν. Δαπανούμε τόσα χρήματα και μετά μου απαντούν οι αρμόδιες αρχές ότι δεν μπορούν να προωθήσουν υποκλοπές. Εγώ μιλούσα για τόνους κοκαίνης που περνάνε σε 11 χώρες του κόσμου και στην ουσία έγινε κατάσκεση 3.000 ε, έγινε κατάσχεση από 3.000 κιλά κοκαίνης και μου λένε ότι δεν μπορούν να γίνουν υποκλοπές. Σας λέω λοιπόν ότι έχω καλύτερη συνεργασία με τους Κολομβιανούς και με τους Ισπανούς, αλλά όχι με ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό μπορώ να σας το τεκμηριώσω. Όταν λήξει η έρευνα θα σας το αποδείξω αυτό. Ελέγχθη ότι τα ναρκωτικά ε, φτάνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια. Δυστυχώς τα αρνητικά στοιχεία δεν είναι πάντα σωστά, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε να τα ερμηνεύσουμε σωστά. Γιατί σε συγκεκριμένα λιμάνια γίνονται κατασχέσεις, γιατί εργαζόμαστε σε αυτά τα λιμάνια. Όμως οι μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης φτάνουν στο Άμστερνταμ, Ρότερνταμ και Αμβέρσας, στις ακτές της Ισπανίας. Εγώ βρέθηκα στο, στην Ουάσιγκτον όπου προέβην σε ανακρίσεις των Μανκούζο που έχουν ε, πατέρα Ιταλό και μητέρα Κολομβιανή, όπου μου είπανε εμείς δεν μπήκαμε από το Γιβραλτάρ, διότι η Μεσόγειος είναι η πιο ασφαλής θάλασσα του κόσμου. Ελέγχεται από τους Ιταλούς και τους Γάλλους. Μου είπαν λοιπόν οι Μανκούζο ότι φέρνουν την κοκαίνη σε ένα μήνυ. Φτάσανε 51 εμπορεύματα στην Ισπανία, στο βορρά της Ισπανίας. Και εκεί δεν έγινε κατάσχεση ούτε μίας παρτίδας. Και αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Όταν βρέθηκα στο Ρότερνταμ είπα στον Γενικό Εισαγγελέα πώς έχουν τα πράγματα. Μετά από παρακολούθηση είδα ότι ο υποέλεγχο έπρεπε να πάει στο Ρότερνταμ για ένα εμπόρευμα το κυβότιο. Δυστυχώς στην Ολλανδία δεν μπορεί να γίνει ετεροχρονισμένη κατάσχεση Φάνηκε λοιπόν ότι αυτό το πρόσωπο είχε δύο κιλά κοκαίνη στο σπίτι του. Μου είπε λοιπόν πρέπει αυτή τη στιγμή να τον συλλάβω γιατί μετά δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί στην Ολλανδία να γίνει ε, ετεροχρονισμένη κατάσχεση ή ε, φυλάκιση, κάτι το οποίο γίνεται στην Ιταλία. Δεν μπορεί να γίνει όμως στην Ολλανδία, στην Ισπανία και στη Γερμανία. Άρα ή θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα γίνει μία ομογενοποίηση αυτών των προδιαγραφών, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, γιατί μιλάμε για διεθνές εμπόριο κοκαίνης. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να ε, ετεροχρονίσουμε, δηλαδή να κατασχέσουμε εκ των υστέρων, επειδή υπάρχουν δύο κιλά κοκαΐνης στο σπίτι και να μην μπορέσουμε να κατασχέσουμε ολόκληρες παρτίδες. γιατί υπάρχει η νοτροπία της πρώην Ανατολικής ε, Γερμανίας, όπου ε, υπήρχε ο φραγκισμός, ε, δηλαδή έπρεπε κανείς να δράσει τάχιστα. Υπάρχουν δηλαδή πολιτισμικές ανασχέσεις. Η Ευρώπη έχει πολλές μαφίες το 2013. Γίνεται ανακύκλωση, αγοράζουν οτιδήποτε. Άμα πάτε στο κέντρο του Λονδίνου, θα δείτε ότι το χειρότερο αυτοκίνητο είναι μία BMW ε, 500. Γιατί αυτό στο κέντρο του Λονδίνου, γιατί δεν υπάρχουν προδιαγραφές καταπολέμησης της ανακύκλωσης του βρώμικου χρήματος στο Λονδίνο. Άκουσα σε μία διάσκεψη ότι στο Λονδίνο δεν φτάνει βρώμικο χρήμα. Δηλαδή, εμείς τι λέμε. Λέμε ότι μερικές πράξεις δεν είναι κατακριτές. Μιλάμε για ενία Ευρώπη όμως. Άρα, θέλω να πω ότι ή θα θεωρήσουμε ότι πρόκειται για εγκληματικές δραστηριότητες που υπάρχουν παντού, γιατί το δικό μας σύστημα είναι το πιο προηγμένο, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δική μας καταπολέμηση της μαφίας. Βεβαίως, ως προς την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω με τη συνθήκη του Προυν. Αλλά οι γνώσεις μας είναι πολύ καλές ως προς την πρόληψη, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, όπου κινηθήκαμε πέρα από τη δράση των αστυνομικών αρχών. Εμείς δεν πρόθουμε τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Η Ντράγκετα κάνει επενδύσεις στην Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, παντού. Αγοράζει ό,τι πωλείται. Αυτό κάνει η ελίτ της μαφίας. Δεν θέλει να πλουτίσει, αλλά να δικαιολογήσει τον πλούτο. Στην Ποκοτά όπου βρισκόμουν ένα μήνα πριν, είδα ότι τα χρήματα δεν καταμετρώνται. Τα βάζουμε στο ζύγι και με αυτά τα χρήματα αγοράζεται ολόκληρος ο κόσμος ε, της Δύσης. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο Γιούργεν Ροτ αυτού του κλάστερ. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, μετά το Duisburg και τους φόνους υπήρξε μεγάλη απήχηση στην δημοσιότητα διότι ήταν όπως σας εξηγήθηκε έξι τα θύματα δηλαδή χύθηκε αίμα και υπήρξαν και πολιτικές αντιδράσεις οι οποίες στράφηκαν γύρω από το θέμα της Ιταλικής μαφίας εν προκειμένου, της Ντράνγκετα και σχετικά βραχυπρόθεσμα υπήρξαν αντιδράσεις διότι το πρόβλημα της Ιταλικής μαφίας στη Γερμανία είναι βέβαια γνωστό από πολλά χρόνια. Οι αστυνομικές υπηρεσίες, είτε ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία ή και ορισμένων ομόσπονδων χωρών, κρατηδίων, γνώριζαν βεβαίω και είχαν ασχοληθεί με την Ιταλική μαφία προηγουμένω. Εγώ εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. Έχω λοιπόν μια επισκόπηση και σχετικά με το τι έχει γίνει στη Γερμανία. Και αυτό μάλιστα σε επίπεδο ομοσπονδιακών κρατηδίων είναι διαφορετικό. Ανά περίπτωση υπάρχουν ορισμένα ομοσπονδιακά κρατήδια όπου ο αγώνας κατά της ε, οργανωμένης εγκληματικότητας και κατά της Ιταλικής μαφίας παίζουν σημαντικό ρόλο, για παράδειγμα Βαβαρία. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι σε άλλα ομόσπονδα κρατήδια, ιδίως τα νέα ομόσπονδα κρατήδια, η Ιταλική μαφία μέχρι τώρα αγνοείται. Για παράδειγμα, Τίριγεν και Σαξονία, δύο σημαντικά ομόσπονα κρατήδια, όπου δραστηριοποιούνται ιδίω οι συμμορίε ε, που προέρχονται από το Σαν Λούκα, στο Έρφουρτ για παράδειγμα, στο Τίριγγεν στην πόλη Έρφουρτ και στη Λιψία και Δρέσδη σε ό,τι αφορά την Σαξονία. Γνωρίζω από τις περιφερειακές αστυνομικές διευθύνσεις από εκθέσεις του 2009 και 10 που αφορούν την Τράγκεντα και την Κοζανόστρα και την Ούνιτα και Καμόρα στην Σαξονία στο Ομοσπονδιακό Κρατήριο της Σαξονίας. Συχνά συμπίπτουν τα συμπεράσματα που συλλέγουν οι διάφορες αυτές οι ε, υπηρεσίες. Μετά από τους φόνους στο Duisburg αυτό τέθηκε ως θέμα και στην Περιφερειακή Βουλή της Αξονίας. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υποστηρίζουν ορισμένοι ότι δεν υπάρχει ιταλική ε, μαφία στην Σαξονία. Στο Τύριγγεν, Θηρίγγι, η κατάσταση είναι παρόμοια. Αρχές της δεκαετίας του 90 δεν υπήρχαν καν ιταλικά εστιατόρια και οι πρώτοι που ήλθαν ήταν οι εκπρόσωποι ε, μιας οικογένειας Σαν Λούκα, ενός κλάν δηλαδή. Πριν αυτά τα είχαμε δει στο Σάρλαντ, άλλο ομοσπονδιακό κρατήδιο, όπου είχαν δραστηριοποιηθεί στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αυτοί λοιπόν άνοιξαν πρώτη Ιταλικά εστιατόρια και μάλιστα σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης και όπου πήγαινε και ο πρωθυπουργός μας και έτρωγε παρόλο που τον είχαν προειδοποιήσει οι ε, αστυνομικοί διευθυντές να μην πηγαίνει σε αυτό το εστιατόριο. Τώρα, το πρόσωπο αυτό που άνοιξε τα πρώτα τελικά εστιατόρια είναι από τους πιο σεβαστούς ε, επιχειρηματίες παρόλο που υπήρχε ήδη, υπήρχαν ήδη πληροφορίες από το 1995 96 ότι το πρόσωπο αυτό είχε πολύ στενές διασυνδέσεις με ιταλικές εγκληματικές οργανώσεις. Έχουμε και άλλη περίπτωση. Άρα αυτά δεν ισχύουν συνολικά για όλη την Γερμανία υπάρχουν επιμέρους ομοσπονδιακά κρατήρια και πόλεις όπου οι οργανώσεις αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο. Ίσως να θυμάστε το 1993, εγώ τουλάχιστον είχα πει τότε σε μια συνδιάσκεψη, είχα μιλήσει για την διασύνδεση της Ιταλικής Μαφίας και της πολιτικής. Είχα τότε πληροφορίες, γιατί είχα συνομιλήσει με ορισμένους πεντήτη, ότι ο τότε επικεφαλής της γερμανικής Τσεντεού είχε φιλικές σχέσεις με έναν Μάριο Λαβοράτο, γνωστή προσωπικότητα στην Τράγκετα, γιατί προέρχεται από μια ε, συγκεκριμένη περιοχή της Καλαβρίας, επίσης εκεί υπήρχε η συμμορία του Φαραώ, ήταν γνωστά τα πράγματα αυτά. Και ωστόσο πέρασε πολύ καιρό μέχρι ότου η αστυνομία και βεβαίως η Ιταλική εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα συλλήψεως, επρόκειτο για σε, μεγάλο, σε μεγάλη έκταση ε, νομοποίηση ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή πλήσιμο βρώμικου χρήματος και ο τότε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Τσεντεού, που σήμερα είναι μάλιστα επίτροπος, έλαβε τις αποστάσεις του από το πρόσωπο αυτό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο κύριος Μάριο Λαβοράτο, που επρόκειτο να καταδικαστεί στην Καλαβρία, μάλιστα κρατήθηκε, προφυλακίστηκε κιόλα και μάλιστα για διάρκεια δύο ετών, αλλά τελικά απελήθη διότι δεν υπήρξαν ε, επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του. Διαθέτει τώρα διάφορα εστιατόρια και στην Φραγκφούρτη και μάλιστα με μαγείρους από τους Φάντα που φαίνεται ότι είναι οι καλύτεροι, οφείλω να το πω αυτό, όπου εκεί πηγαίνει και τρώει η πραγματική αριστοκρατία της Φραγκφούρτης και μάλιστα θα δείτε και στους τοίχους ε, του ε, εστιατορίου φωτογραφίες ε, υψηλά ισταμένων και το εστιατόριο αυτό ανήκει, το εστιατόριο αυτό ανήκει σε ανιψιό του Μάριο Λαβαράτο, ο οποίος λέει ότι εγώ και μετά μάλιστα από την κράτησή μου ανέβηκα και κοινωνικά. Το βγαίνει και βγαίνει και το λέει ο ίδιος. Η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση έχει ασχοληθεί και με την Ιταλική μαφία, ωστόσο το προσωπικό της έχει μειωθεί. Δεν έχει τους πόρους ούτε οικονομικά ούτε απόψεις τελεχώσεως για να ασχοληθεί με το είδος αυτό της εγκληματικότητας. Τα ίδια θα δείτε αν πάτε και σε άλλο ομοσπονδιακό κρατήδιο, Mecklenburg, Mecklenburg Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 φαινόταν καθαρά ότι η Σάκρα Κορώνα Ούνιτα, άλλη εγκληματική οργάνωση, δραστηριοποιούνταν και επένδυε σε ξενοδοχεία και εστιατόρια στην ακτή της ε, Βαλτικής. Αυτοί όλοι έχουν επαφές με την Ιταλία. Όμως δεν επετράπει στην εισαγγελία να ε, ερευνήσει περισσότερο διότι δεν διέθετε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και πόρους προσωπικού για να κάνει περισσότερες έρευνες. Αν πάτε τώρα στην πόλη Μπίνς θα δείτε ότι βεβαίω όλα αυτά τα εστιατόρια και ταβέρνε κτλ. είναι απολύτω νόμιμα και οι αστυνομικέ αρχέ δεν έχουν πλέον απολύτω καμία δυνατότητα να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση. Ωστόσο, η συνειδητοποίηση στην πολιτική ελίτ είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν μιλεί κανεί στη Γερμανία για εγκληματικέ οργανώσει, δεν υπάρχει απολύτω καμία συνείδηση μεταξύ των πολιτικών ότι η οργανωμένη μαφία μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για τη δημοκρατία. Βλέπετε σε διοργανώσεις και ο Κατέρη θα σας το επιβεβαιώσει, όταν πρόκειται για οργανωμένη εγκληματικότητα δεν βλέπετε ποτέ κάποιον πολιτικό που να έρθει να ενημερωθεί. Ούτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ούτε σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν βλέπετε ποτέ πολιτικό που να έρθει να ασχοληθεί επί μακρόν με την οργανωμένη εγκληματικότητα. Στη Γερμανία, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο και νομίζω τα ξέρω αρκετά καλά τα πράγματα. Στην Ιταλία σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Επομένω, η συνειδητοποίηση είναι εντελώ στο περίπου. Υπάρχει έκθεση τη Εγκληματολογική Υπηρεσία από το 2006 που ασχολείται εκτεταμένα με την Τράγκετα. Ε, ε, περιγράφει τον κίνδυνο, αναφέρει για τη διασυνδέση με την Ιταλία. Ούτε μια λέξη ωστόσο δεν λέει για την επιρροή της δράγκετα στην Γερμανία. Ότι αγοράζει τα ταμιευτήρια και τράπεζες στη Ρουμανία, αυτά τα λέει. Στη Γερμανία, για τη Γερμανία δεν λέει τίποτα η έκθεση αυτή. Το πρόβλημα, όπως το εξήγησε ο κ. Γέγκερ προηγουμένως και ο κ. Κρατέρη ούτως ή άλλως τα λέει αυτά εδώ και καιρό, το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ ότι η αστυνομία δεν θέλει να αντιμετωπίσει την εγκληματική αυτή δραστηριότητα, αλλά η, ε, αστυνομία δεν έχει επαρκή κάλυψη από την πολιτική για να διεξαγάγει τον αγώνα αυτό. Αν παρακολουθήσετε τις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της αστυνομίας τα τελευταια δυο δύο-τρία χρόνια, θα δείτε καταρχήν μείωση των θέσεων προσωπικού ε, που καταπολεμά την οργανωμένη εγκληματικότητα λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης. Για παράδειγμα, εκεί όπου χρειάζονται διερμηνείς, περικοπές. Επομένως, δεν είναι δυνατόν πλέον να γίνουν οι έρευνες. Υπάρχουν ίσως κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά όλοι οι εγκληματολόγοι στη Γερμανία θα σας πούν υπάρχει ίσως και κάποια ε, περίπτωση όπου γίνονται κάποιες επενδύσεις, για παράδειγμα στη Φραγκφούρτη από την οποία προέρχομαι, τμήματα των ακινήτων που αγοράζονται τώρα αγοράζονται από μια ε, ομάδα από τη Τζένοβα και υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μελών της Δράγκεντα με μέλη της Κοζανόστρα και με Γερμανούς δικηγόρους. Εγώ αυτά τα στοιχεία τα έθεσα υπόψη της αστυνομίας της Φραγκφούρτης και η απάντηση ήταν ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα να διαρευνήσουμε. Άλλο θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό και ο κύριος Γέγκερ επίσης το έθιξε η στόχευση μονάχα στην Ιταλική μαφία είναι λάθος. Στη Γερμανία έχουμε και άλλες εγκληματικές οργανώσεις με πολύ μεγάλη επιρροή. Ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό, η, η αλβανική μαφία παίζει κέριο ρόλο και στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και, στο, ε, και στη σωματεμπορία και στους εκβιασμούς. Ένας γερουσιαστής, σκεφτείτε, ο Ρόλαν Σίδλ, γερμανικού ε, κρατηδίου που ήταν γερουσιαστές Διαουσιαστή αρμόδιος για τα εσωτερικά και γραμματέας του Υπουργείου του ήταν δικηγόρος ο οποίος εκπροσωπούσε τους μεγαλύτερους μαφιόζους στη Γερμανία. Αυτός λοιπόν υποστηρίχτηκε από τους λεγόμενους αδελφούς Οσμάνι. Αυτοί οι αδελφοί Οσμάνι ανήκουν στην οικογένεια Οσμάνι από, τους, από τις πιο σημαντικές οικογένειες, αλβανικές οικογένειες, εγκληματικές οικογένειες δηλαδή, που είχαν μεγάλη επιρροή στο Σαν Πάουλι, στο, στη Βόρεια Γερμανία. Αυτοί ασχολήθηκαν με κοκαίνη και με πολύ νεαρά κορίτσια. Αυτά τα πράγματα βγήκαν, σκεφτείτε τώρα υπήρχε μάλιστα τότε κυβερνούσε συνασπισμός με την Τσεντεού στο Αμβούργο. Μετά όταν αυτός ο γερουσιαστής Σίτλ ε, εμφανίστηκε ως ομοφιλόφιλος, αυτό οδήγησε σε μια ρήξη στο συνασπισμό. Μέχρι τότε ωστόσο είχαν αποτραπεί οποιασδήποτε έρευνες. Παρετήθηκαν ε, αστυνομικοί διευθυντές διότι αυτό το πρόσωπο, αυτός ο ε, Σίδλ, είχε γίνει γεροστιαστής αρμόδιος για τα εσωτερικά, δηλαδή ένα είδος υπουργών εσωτερικών στην περιφερειακή αυτή κυβέρνηση. Για να ολοκληρώσω, έχουμε τελείως διαφορετικές διαστάσεις Έχουμε τώρα τις κοινοπραξίες μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, εταιριών με γερμανικές επιχειρήσεις. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο, που δεν αφορά μονάχα την Ιταλία αλλά την Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία είναι γνωστό ότι τη μεγαλύτερη επιρροή έχει η εγκληματική ομάδα TIM που είναι αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, είναι πραγματική αυτοκρατορία η ομάδα Team. Ξεκίνησαν έρευνες οι οποίες παρεμποδίστηκαν. Υπάρχουν δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη. Εγώ ο ίδιος μίλησα με τον Κάμινοφ για τις κατηγορίες καταγγελίες αυτές. Ε, η οργάνωση αυτή προβαίνει σε φόνους εκβιασμούς. Αυτός είναι άνθρωπος αφελής. Το ότι ε, διευθύνει ολόκληρη επιχείρηση δισεκατομμυρίων, αλλά αυτό είναι βουλγαρικό πρόβλημα. Πρέπει να το λύσει η Βουλγαρία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η επιχείρηση ξεκινά τώρα κοινοπραξίες με γερμανικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα την Fraport, την ε, ε, εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Άρα, εγκληματικές οργανώσεις μπαίνουν σε επιχειρήσεις με γερμανικές ή άλλες μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις. Μιλώ για joint ventures, όπου εκεί παίζουν βέβαια κέριο ρόλο και τα οικονομικά συμφέροντα και τα πολιτικά συμφέροντα. Αυτό να αγωνιστεί κανείς κατά τέτοιων ε, δράσεων θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως σας είπα εγώ παρακολουθώ τα πράγματα αυτά εδώ και μια τριακονταετία και βλέπω ότι τα πράγματα δεν γίνονται καλύτερα αλλά μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης γίνεται όλο και δυσκολότερο για τις δημοκρατικές χώρες να καταπολεμήσουν αυτή την εγκληματικότητα, διότι η διαδικτύωση μεταξύ παρανομίας και νομιμότητας γίνεται όλο και πιο στενή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νιούτον Ντάν ζήτησε το λόγο μέσα στα πλαίσια της συζήτησης μόλις, μόλις αρχίζει. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικές ε, και οι τρεις παρουσιάσεις. Ε, λυπάμαι που έχουμε τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να μας δώσετε τις ε, παρουσιάσεις σας έτσι ώστε να τις μελετήσουμε. Προς τον ε, Γερμανό ε, συνάδελφο που μίλησε πρώτος, τον κύριο Γέγκερ, θα ήθελα να υποβάλω την εξής ερώτηση. Εάν κατάλαβα καλά, μιλήσατε για εναρμόνιση των κανόνων των 28 κρατών μελών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό να υπάρχει μία ευρωπαϊκή FBI που να μπορέσει να δράσει ομοσπονδιακά. Ε, περιλαμβάνω και την Κροατία, η οποία θα προσχωρήσει σε λίγες μέρες. Πρόκειται για ένα Ηράκλειο έργο. Δεν θα το τελειώσουμε ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία υπηρεσία τύπου FBI, δηλαδή να λάβουμε υπόψη ότι αυτές οι ομάδες είναι διεθνείς. Άρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα αστυνόμευσης που να έχει τον ίδιο χαρακτήρα. Δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε γιατί είναι πολιτική ερώτηση και εσείς ε, είστε αστυνομικές αρχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Ευρώπη είναι τόσο φαραλέα ώστε να δώσει μάχη σε αυτό το επίπεδο. Γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμήσουμε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Πρόκειται για μια πολιτική δήλωση που ίσως δεν θέλετε να κάνετε. Προς τον Ιταλό συνάδελφο, προς τον κύριο Γκρατέρη, θα ήθελα να υποβάλω την εξή ερώτηση. Η εισαγωγή κοκαΐνης, ξέρω ότι έχετε δίκιο, έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το θέμα στις εισαγωγές είναι πώς να ελέγξουμε αυτά τα κάργο. Μερικοί από εμά τη είπα λίγες εβδομάδες πριν, είδαμε πώς ε, το αντιμετωπίζουμε. Πήγαμε στο λιμάνι της ε, Νέας Υόρκης και είδαμε τα μεγάλα κοντέινερ να φτάνουν. Οι αστυνομικές αρχές μας εξήγησαν τι συμβαίνει και μας είπε «Μπορώ να ελέγξω μόνο το 5% των εμπορευματοκιβωτίων που μπαίνουν» και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κοκαίνη από την Καραϊβική και άλλα εμπορεύματα. Λέω τότε γιατί δεν έλεγχετε τα άλλα. Λέει γιατί ο, δήμαρχος της Νέας Υόρκης μου λέει ότι έχουμε Έχουμε σειρά πλοίων που πρέπει να εκφορτώσουν και τα σούπερ μάρκετ λένε τις, μας λένε επίσης ότι θέλουν αυτά τα προϊόντα να φτάσουν σε αυτά. Μας παραπονούνται λοιπόν να μην παρακολύσουμε το εμπόριο. Πώς λοιπόν εμείς στην Αμβέρσα, στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ μπορούμε να ελέγξουμε το κάθε εμπόρευμα το κυβότιο. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα να ακούσω μία λύση αλλά θα καθυστερήσουμε υπερβολικά το ενδοκινοτικό εμπόριο, αν θέλουμε να ελέγξουμε τα πάντα. Δεύτερον, μιλήσατε με μεγάλο πάθος και είπατε ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε το Ιταλικό σύστημα αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι η Ιταλία είναι εξαιρετική κόρα και σας αγαπώ πολύ, αλλά η εικόνα της Ιταλίας και ο ίδιος ο κύριος Μπερλουσκόνη συνέφερε σε αυτό, είναι μία διαφθαρμένη χώρα. Και όταν μας λέτε ότι πρέπει να εισαγάγουμε το Ιταλικό σύστημα, αυτό θα οδηγήσει σε θυμηδία στην Ευρώπη. Τη στιγμή που έχουμε τον κύριο Μπερλουσκόνη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διαφθορά, αλλά δεν έχει φυλακιστεί, Καταλαβαίνετε ότι κανένας μας δεν θέλει να εγκρίνει το Ιταλικό σύστημα. Καταλαβαίνω ότι είσαστε ειλικρινείς και εσείς έχετε ένα καλό σύστημα, αλλά θα πρέπει να περάσει το σύστημά σας παρά την Ιταλική, ε, αυτό το Ιταλικό σήμα, αν θέλετε. Λυπάμαι που μίλησα κατά αυτόν τον τρόπο. Και τρίτον, προς, τους, προς το γερμανό συνάδελφο, νομίζω ότι θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή δεν υπάρχει ενσυνειδητότητα από την πολιτική ελίτ. Και αυτό είναι ο στόχος αυτής της Επιτροπής. Εμείς είμαστε πολιτικοί, όχι ελίτ, απλώς πολιτικοί που προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση ενσυνειδητότητας, ευρύτατης συνειδητοποίησης του θέματος και θέλουμε να πούμε στους πολιτικούς ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν συμβαίνει τίποτα. Εάν μπορέσετε να μας βοηθήσετε με υποδείξεις, εμείς έχουμε προθεσμία για την τελική έκθεση μέχρι το τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί εάν κανείς δεν δώσει σημασία στη, το φθινόπωρο στην έκθεσή μας, τότε ε, δεν θα γίνει τίποτα. Απλώς θα ανήκουν σαμπάνια σε αυτά τα εξαιρετικά ιταλικά εστιατόρια τα οποία προαναφέραμε και τίποτα άλλο δεν θα γίνει. Ευχαριστώ, Μπίλ. Μία διευκρίνηση θέλω να κάνω. Όταν ο συνάδελφος μίλησε για την επιθυμία να υιοθετήσουμε την νομοθεσία αντιμάφια, αναφέρεται σε όλα τα μέτρα, σε όλες τις νομοθεσίες που επέτρεψαν ε, σε μία σειρά από χώρες να έχουν επιτυχίες. Πολύ σωστά τονίζεις το θέμα της αξιοπιστίας μπορεί να έχει μια χώρα όταν διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί δεν κάνουν κάποια πράγματα. Όμως, όπως είπε και ο Αγγελέας, η Ιταλία έχει μια νομοθεσία κατά της διαφθοράς εντελώς αναποτελεσματική. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ε, το θέμα της αξιοπιστίας της Ιταλίας ε, στο στο μέτωπο της ε, καταπολέμησης της ε, μαφιόζικης εγκληματικότητας. Για να δημιουργηθεί αυτή η νομοθεσία ε, κατά της μαφίας πέθαναν εκατοντάδες δικαστές. Και εγώ αισθάνομαι μηχανία και πολλοί άλλοι αισθάνονται μηχανία. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε τα θετικά στοιχεία που έχει η νομοθεσία στη χώρα μου. Ο κύριος Μαστέλα θέλει να πάρει το, το λόγο και ας αφήσουμε και λίγο χρόνο στον δικαστή, για να, στον εισαγγελέα δηλαδή, για να απαντήσει. Εγώ θα, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα με βάση την εμπειρία μου. Προφανώς δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ της Ιταλικής και Γερμανικής νομοθεσίας. Αυτό το επεισόδιο που αναφέρατε των φόνων το Duisburg ακριβώς δείχνει αυτό το, αυτή τη διαφορά. Η Ιταλία είχε δικαστές που συνεργάζονταν με την Γαλλία, με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά όχι με τη Γερμανία. Όπως είπε και ο κύριος Κρατέρη, οι κανόνες δεν ε, συνέπιπταν. Επομένως, ε, υπήρχε πρόβλημα αποτελεσματικότητας ε, για οποιονδήποτε ασχολούνταν με αυτό το κλιματικό φαινόμενο. Αυτό το επεισόδιο μας έδειξε ότι αυτός ο καρκίνος, αυτό το καρκίνωμα το, της Ιταλίας ε, μεταλαμπαδεύτηκε ας πούμε, ε, εμφανίστηκε εν πάση στη Γερμανία. Το φαινόμενο της μαφίας ή της, των μαφιών όπως είπε ο τελευταίος εισηγητής, ε, γιατί δεν υπάρχει ο, μία Ιταλική μαφία. Υπάρχουν πολλές μαφίες που υπάρχουν στην Ευρώπη και ε, υπάρχει ε, διασύνδεση μεταξύ τους σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ένας κατάλληλος νόμος. Πρέπει να συνδέσουμε τις ε, νομοθεσίες αυτές και οι νομοθεσίες αυτές θα πρέπει να συγκλίνουν. Ούτε πρέπει να λέμε ότι κάποιοι, ας πούμε, κάποιες νομοθεσίες είναι θετικές, κάποιες είναι αρνητικές, ούτε πρέπει να πέφτουμε θύματα εθνικών εγωισμών. η Ντράγκετα είχε μπει στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτη. Η Ντράγκετα ε, στον Καναδά, στην Αυστραλία, έτσι και στη Γερμανία, ας πούμε, μπήκε στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτη. όπως είπε και ο καθηγητής ε, Κρατέρη. Και είναι η, μία από τις Ιταλικέ ε, Ιταλικές που παράγει τον περισσότερο πλούτο. Και το βασικό για την Ντράγκετα είναι ότι ήθελε να προωθήσει τα συμφέροντά της. Η Ιταλία προφανώς θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το φαινόμενο. Καταλαβαίνετε ότι είναι Ιταλική ασθένεια αυτή και επομένως ε, έχουμε και τους κατάλληλους γιατρούς. Δεν είναι ότι είμαστε καλύτεροι. Δεν είναι ότι οι ερευνητές μας είναι καλύτεροι. Έγιναν καλύτεροι γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Γιατί αν δεν έχεις τη γνώση, αν δεν... Αν δεν έχεις μάλλον το φαινόμενο, για ποιο λόγο να αποκτήσεις τη γνώση. Το ίδιο συμβαίνει και στην ιατρική μην φανταστείτε ότι είναι θέμα, ας πούμε, ιταλικής α, Εγώ ως υπουργό ε, είχα την τιμή να ε, συναντηθώ με τον πρόεδρο του Μεξικού, να συνεργαστώ με αμερικανικές αρχές, με χώρες Ανατολικής Ευρώπης, ε, που ενδιαφέρονταν να δουν την ομοθέσια που προωθούσε η Ιταλία με σκοπό να αντιμετωπίσει την μαφία. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ποια είναι η γνώμη μου είναι σαφές ότι όταν υπάρχει συνεργασία δίνουμε κίνητρα και στους πολιτικούς να συνεργαστούν μεταξύ τους. Όταν εμείς συνεργαζόμαστε και οι πολιτικοί συνεργάζονται. Αν ε, η Ευρώπη των 27-28 χωρών ε, εργάζεται κάθε χώρα μόνη της, προφανώς παραμένει αναποτελεσματική. Δέστε πώς αντιμετωπίζονται σε άλλες χώρες, ας πούμε, τα προβλήματα των ε, ναρκωτικών. Υπάρχουν κενά στη συνεργασία μας. Ε, πρέπει να, να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη έκλεινε τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο. Θεωρούσε ότι είναι ιταλική, υπόθεση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν ισχύει πια αυτό. Σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, υπάρχει μία ανάμειξη και σε άλλες χώρες. Φυσικά ε, η εγκληματικότητα απλώνει τα πλοκάμια της και οι εγκληματίες ενός κλάδου συνδέονται με εγκληματίες άλλου. Ίσως είναι κασανδρισμός αυτό που θα πω, αλλά εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να δώσουμε ένα πλαίσιο σε όλο αυτό το, φαινόμενο. Ε, οι Ιταλοί δεν μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους, ούτε η Γερμανία από μόνοι τους. Αυτό το φαινόμενο μας αφορά όλους. Και ελπίζω οι νομοθεσίες των διαφόρων χωρών να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Πάντως, έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα αυτά, έχει αλλάξει ο τρόπος που ερευνούμε αυτά τα φαινόμενα και που τα διώκουμε. Ευχαριστώ. Ο κ. Σόντεργαρντ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γέγκερ μίλησε για μια ανταλλαγή πληροφοριών για δακτυλικά αποτυπώματα που ανταλλάχθηκαν κτλ. Είναι σίγουρο ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να διευκολύνουμε την έρευνα, να διευκολύνουμε τον αγώνα κατά της εγκληματικότητας, του εγκλήματος και κυρίως της, του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα να μου πείτε όμως αν υπάρχει κάποια αρνητική πτυχή σε αυτό. Αναφερθήκατε σε μια περιόριστη ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν υπάρχει όριο. Όμως, δεν υπάρχει όριο στις πληροφορίες που μπορούν να ανταλλαγούν. Και γιατί σας θέτω αυτό το ερώτημα. Γιατί είπατε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων αρχών. Αυτό είπατε. Και το ερώτημά μου είναι, υπάρχει βάση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να πετύχουμε αυτή την εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων αρχών. Υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Βλέπετε τι γίνεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ε, πρέπει να, έπρεπε να υιοθετήσουμε μία έκθεση για το σεισμό στην Ακούιλα. Και διαπιστώσαμε ότι συστηματικά οι πληροφορίες που μας δίδονταν από τις ε, Ιταλικές αρχές ήταν λανθασμένες. Υπάρχει λοιπόν, εδώ δημιουργείται και προκύπτει μια δυσπιστία. Θα ήθελα να μου πείτε, οι αρχές λοιπόν ε, έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους ή μήπως υπάρχει ο κίνδυνος ότι η μαφία διεισδύει και βάζει τους δικούς της στις διάφορες αρχές. Φυσικά πρέπει να καταπολεμούμε συστηματικά τις εγκληματικές οργανώσεις. Αλλά αυτή η οργανωμένη εγκληματικότητα, ε, αυτό το οργανωμένο έγκλημα δεν διεισδύει σε διάφορα επίπεδα. Όταν ανταλλάσσουμε ευρέως πληροφορίες, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στις ε, εγκληματικές οργανώσεις να αποκτήσουν όπλα. Δεν διαραίουν κάποια από τα στοιχεία σε αυτές τις οργανώσεις. δεν θα έπρεπε να έχουμε κάποιο περιορισμό στην ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αστυνομικών αρχών Φερρυπίν. Κυρίες, κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Κρατέρη. Είπατε ότι δεν έχετε αρκετούς πόρους για να ασχοληθείτε με τα μεγάλα φαινόμενα εγκληματικότητας. Είπατε ότι οι χώρες δεν έχουν αυτές, αυτούς τους πόρους. Ε, εάν επρόκειτο για τη Δανία, θα έθετα το ερώτημα στη Δανία αλλά μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποια είναι αυτή η χώρα που δεν έχει τους απαραίτητους πόρους. Μπορείτε να την ονομάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπορσελίνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι από αυτή την άκρο ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, ανακύπτει το θέμα της ανάγκης μιας μεγαλύτερης Ευρώπης, ε, δηλαδή συστήματα έρευνας, διερεύνησης, ε, δικαστικής αρρωγής και ούτω καθεξής. Αυτά μας οδήγησαν και στη σύσταση αυτής της Επιτροπής. Η Επιτροπή Κρίμη υπάρχει διότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να κάνουμε κάτι περισσότερο. Αυτό είναι ύψης της σημασίας. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι μέσα ήδη διαθέταμε, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσαμε ή δεν τα χρησιμοποιούσαμε σωστά. Γι' αυτό μιλήσαμε για κοινέ ερευνητικές επιτροπές. Ε, δεν υπάρχουν κονδύλια βεβαίως, δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων αλλά επαναλαμβάνω ότι το κανονιστικό πλαίσιο προϋπήρχε για τη συνεργασία αυτή, που όμως στην πράξη δεν ίσχυσε. Στην Ιταλία υπάρχουν πολλά ε, ελλείμματα, αλλά είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες και πιο ισχυρές μαφίες γεννήθηκαν στην Ιταλία. Αυτό το γνωρίζουμε και γι' αυτό έχουμε πλήρη επίγνωση του εγχειρήματος και γι' αυτό η Ιταλία διέθετε τα κατάλληλα μέσα νωρίτερα, πιο έγκαιρα. Οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούσαν να δράσουν στη Γερμανία γιατί δεν έχουν ε, πολιτική κάλυψη, ενώ στην Ιταλία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το Ιταλικό σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή διακρίνουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το δικό μας σύστημα μπορεί να προκαλέσει θυμηδία και υπάρχουν ελλείψεις, αλλά σε σχέση με το Duisburg και ό,τι συνέβη, θα ήθελα να καταλάβω το εξής. Η Ιταλική μαφία είναι υπεύθυνη για τη σφαγή του Duisburg. Δηλαδή υπάρχει μόνο η Ιταλική μαφία στη Γερμανία ή δρά η Ιταλική μαφία και στη Γερμανία και άρχισε να πλουτίζει στη Γερμανία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει συνεργασία με Ολλανδούς, Γερμανούς, Γάλλους και ούτω καθεξής. Διότι αυτός ο πλουτισμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνεργασία. Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι δυνατότητες που ε, υπάρχουν και πόσο είναι υπεύθυνη, τι ευθύνες φέρει η χώρα που φιλοξενεί για αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί είναι πολύ απλουστευτικό αν λέμε ότι οι Ιταλοί, οι μαφιόζοι ε, κάνουν τα εγκλήματα και μετά πλουτίζουν στο εξωτερικό. Μα πώς γίνεται αυτός ο πλουτισμός σε μια άλλη χώρα και και ποια ευθύνη φέρει η Ευρώπη σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο κύριος Καρόνα έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να πω τα εξής που αφορά εμάς τα μέλη αυτής της Επιτροπής πολύ περισσότερο από τους προσκεκλημένους μας και μετά θα κάνω τις ερωτήσεις μου. Εμείς θα πρέπει στην εργασία μας αυτή να λάβουμε υπόψη ένα συγκεκριμένο στοιχείο, ένα δεδομένο. Δηλαδή, οι εγκληματικές οργανώσεις δεν αφορούν μόνο ορισμένες χώρες και περιφέρειες. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά και τα 27 κράτη-μέλη και ιδιαίτερα ορισμένες χώρες. Με, με προεξάρχουσα την Ελβετία που δεν, είναι στην Ευρωπαϊκή, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τραπεζικά οικονομικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της σκέψης μας. Και αυτό σας το λέω γιατί προέρχομαι από μία συγκεκριμένη περιφέρεια. Εγώ προέρχομαι από την Εμίλια Ρωμάνια, η οποία είχε την εντύπωση ότι δεν συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία της οικονομικής διείσδυσης των εγκληματικών οργανώσεων. Ζούσε αυτή τη φενάκη δηλαδή, μαζί με άλλες περιφέρειες του βορρά της Ευρώπης. Μετά όμως είδε ότι δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποια μέρα ξύπνησε και είδε ότι πολλοί οικονομικοί τομείς έχουν εμπλακεί και βρίσκονται υπό τον έλεγχο εγκληματικών οργανώσεων και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ωραίο. και αυτό το λέω αναφερόμενος σε αυτά που προείπε ο δόκτωρ Ροτ. Δηλαδή, πολλές χώρες του βορρά της Ευρώπης ίσως αυταπατώνται και πιστεύουν ότι οι εγκληματικές οργανώσεις ιταλικής προέλευσης ή μη δεν έχουν καμία σχέση με αυτές, ενώ στην ουσία ελέγχουν μεγάλα τμήματα του οικονομικού ιστού. Γι' αυτό και νομίζω ότι έπρεπε να πω αυτές τις σκέψεις. Μετά θα τις δούμε ε, μέσα στα πλαίσια της έκθεσης του κυρίου Γιακολίνο. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου για να μπορέσουμε να δώσουμε μία ολοκληρωμένη απάντηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γέγκερ τα εξή. Ε, μετά τη σφαγή του Ντόισμπουργκ, η γερμανική κοινή γνώμη αντέδρασε και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η φαιά ζώνη πώς ορίζεται. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση των εγκληματικών οργανώσεων και του εμπορικού τομέα ή μάλλον των συμβολεογράφων, δικηγόρων κλπ. κλπ που αποτελούν το επίκεντρο δραστηριότητας, δηλαδή ε, αποτελούν διάβλο δραστηριότητας των εγκληματικών οργανώσεων. Πώς είναι η κατάσταση. Προς τον δόκτορα Γκρατέρη θα ήθελα να αποβάλω την εξής ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα και με βάση τη δική σας πείρα, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ξέρετε ότι υπάρχει, υπάρχουν διστάμενες απόψεις ως προς τις υποκλοπές. Άκουσα και τις διάφορες επικρίσεις που ακούστηκαν ότι δεν έχουμε μία σωστή τράπεζα δεδομένων ανείχνευσης DNA. Εμείς ως Ιταλοί Πού θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί τα επόμενα χρόνια για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δίας Δεμέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη διότι έπρεπε να βρεθώ αλλού ε, καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, δηλαδή βρέθηκα ε, σε επιτροπές που ασχολήθηκαν με διάφορα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε μία δυναμική σε αυτή τη συζήτηση και στα θέματα που μας απασχολούν. Εκτιμώ ιδιαίτερα ε, το ενδιαφέρον του κυρίου Νιούτον Ταν ο οποίος μίλησε για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής FBI. Νομίζει ότι αυτή θα ήταν πανάκια, εγώ όχι. Πιστεύω ότι μία υπηρεσία τύπου FBI έχει μία ομοσπονδιακή ε, μορφή μιας μεγάλης ε, δημοκρατικής χώρας, ε, η οποία έχει και μεγάλες βαλωτότητες. Δηλαδή υπάρχει η FBI αλλά εκεί ε, ξεπλένεται και, με το, και το μεγαλύτερο τμήμα του χρήματος. Εκεί υπάρχει η περισσότερη κοκαίνη και διακινείται. Εκεί γίνεται η μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή στη ΣΥΠΑ, όπου υπάρχει και η FBI. Γι' αυτό η Ευρώπη καταρχήν δεν φέρει ομοσπονδιακή μορφή και πολιτικά. Δεν μπορεί να κινηθεί προς μία υπηρεσία τύπου FBI και δεν θα ήταν και λύση αυτή. Σε επίπεδο ασφάλειας μπορεί να ανακύψουν και πολιτικά ζητήματα, αλλά δεν υπάρχουν απόλυτες απαντήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Διότι φιλοσοφικά και υλικά δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια πουθενά. Πιστεύω ειλικρινά, για να μπω στην ουσία αυτής της συζήτησης, είναι αδύνατο να ελέγξουμε όλα τα εμπορευματοκιβώτια που μπαίνουν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και δεν μπορούν να ελέγχουν δεν μπορεί να ελεγχθεί το διαμετακομιστικό αυτό εμπόριο ούτε στη δική μου χώρα, ούτε στα δικά μας λιμάνια από όπου προέρχονται τα εμπορεύματα της Βορείου Αφρικής. Και αυτό αφορά και το στενό του ε, Γιβραλτάρ. Ξέρετε ε, ότι υπάρχει μεγάλο εμπόριο μεταξύ των βορείων ακτών της Αφρικής και της Ευρώπης. Ως προς την Ιταλία και το σύστημα ασφάλειας. Η Ιταλία έχει θεσμοθετήσει αυτό το τομέα, γι' αυτό και έχει όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να ελέγξει αυτό το τομέα ε, όταν υπάρχουν εγκληματικές δραστηριότητες ή απαρχή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πιστεύω ότι η Ιταλία με αυτή την ισχυρή, ισχυρή θεσμοθέτηση έχει ελέγξει το τομέα και το γνωρίζω εξιδίων γιατί συνεργάστηκα σε θέματα ασφαλείας με τις Ιταλικές αρχές με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στην ε, ε, υπόθεση Ντιτζενάρο ιδιαίτερα. Γι' αυτό και υποστηρίζω τους ε, Μαστέλα, ε, Μπορσελίνο και Κατόρνα. επειδή όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ ιδεατού και πραγματικού, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι αδύνατο να καταπολεμήσουμε το έγκλημα σε όλες τις διαστάσεις του. Δηλαδή, ας δούμε και αυτούς που κινούνται αυτόνομα. Ε, στις, ε, ε, ε, έχουν επιτεθεί στη Βοστόνη, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Πώς θα τους καταπολεμήσουμε. Δηλαδή, ο Ζιλ Ντε Κέρκοπ υπέβαλε μία έκθεση για να μιλήσει για τη διάσταση αυτού του φαινομένου και να μιλήσει για τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα και τα δεδομένα που θα μπορούσαμε να έχουμε σε επίπεδο ασφάλειας εθνικής και ευρωπαϊκής. Τώρα, ως προς την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ενισχυθεί. ή διμερείς είναι εύκολη. Όταν είναι πολυμερής όμως και αφορά θέματα ασφαλείας δεν είναι εύκολη, όπως ξέρει και η Πρόεδρός μας. Όπου είδαμε και τη συνεργασία μεταξύ των Καραμπινιέρη και της Guardia Civil της Ισπανίας με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε και την υποδομή της Europol και βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες και πρόοδος σε αυτό το τομέα. μετά από την προσεχή έγκριση του νέου κανονισμού της ε, Europol που θα εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι η Europol θα έχει ενισχυμένες δομές και θα υπάρχει μεγαλύτερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσα στα πλαίσια της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Αυτά θα ήθελα να πω με βάση και τη δική μου πείρα. Γιατί υπάρχουν δύο πλευρές του νομίσματος, αλλά εγώ τάσομαι υπέρ της ασφάλειας πρωτίστως. Ευχαριστώ, Αγκουστίν. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους συγγητές για να απαντήσουν και να κάνω και κάποιες... Ε, ε, να δώσουν και κάποιες διευκρινήσεις. είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες με κάποιους συναδέλφους που εκπροσωπούσαν άλλα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Υποστηρίζοντας όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής, ότι υπάρχει και η πολιτική διάσταση της λύσης του προβλήματος. Ε, θέλω να πω ότι για το θέμα που μας απασχολεί, Δεν ήθελα να στείλω mail στους συναδέλφους που ανήκουν στο συγκεκριμένο ε, κράτος μέλος, mail μεταφρασμένο στη γλώσσα τους για να συμμετάσχουν στη σημερινή συζήτηση. Ε, γιατί ήξερα ότι οι ομιλητές μας δεν θα μας απογοήτευαν. Δηλαδή, θα, αναφερό, θα αναφερόντουσαν σε όλα αυτά τα προβλήματα, στην αρμόνιση των δικαστικών συστημάτων, ε, στα ερευνητικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες. Μιλάω λοιπόν για αυτή τη συγκεκριμένη χώρα και για, τους, και για τα άτομα που προέρχονται από αυτή την χώρα. Η απουσία των συναδέλφων από αυτή τη χώρα είναι πολύ σημαντική ε, για μένα. Γιατί τελικά δεν θέλουν να καταλάβουν. Ζητώ συγγνώμη για, για τον τρόπο που μιλάω. Έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα. Προσπαθούμε να τα δρομολογήσουμε. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο κτλ. Αλλά αντιμετωπίζουμε διάφορα εμπόδια που μπορεί να είναι πολιτικής ιδεολογικής φύσεως. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι δράσεις που προωθούνται ε, υποκινούνται από τις κυβερνήσεις των, αυτών των κρατών από τα οποία προέρχονται αυτοί οι συνάδελφοι. Όταν παρουσιαστεί η έκθεση της, του συναδέλφου Γιακολίνο, πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί στη συζήτησή μας. Γιατί αλλιώς θα πούμε διάφορα πράγματα, χωρίς όμως δύναμη, χωρίς ισχύ, χωρίς θένος και χωρίς να προωθήσουμε τα μέτρα τα οποία πραγματικά πρέπει να εφαρμοστούν. Με τον Αγκουστίν τις προηγούμενες μέρες ανταλλάξαμε διάφορα mail για διάφορες έρευνες που κάνουν από κοινού Ιταλικές και Ισπανικές αρχές. Ε, και ακριβώς αυτό δείχνει την καλή σχέση που έχουν οι αρχές. Ο εισαγγελέα, ο κύριος Κρατέρη, είπε ότι κατάφερε να δημιουργήσει προσωπικές σχέσεις με τους ομολόγους του σε διάφορα κράτη-μέλη, ακόμα και σε τρίτες χώρες. Αλλά οι προσωπικές σχέσεις δεν είναι η μόνη λύση. Εμείς πρέπει να θέσουμε τις βάσεις, ούτως ώστε να φτάσουμε σε εναρμόνιση των δικαστικών συστημάτων. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες από χώρα σε χώρα και με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και του αποδίδουμε διαφορετικό βαθμό απειλής. Συμφωνώ με τον Αγκουστίν ότι χρειαζόμαστε και υποστήριξη και την υποστήριξη της Europol, αλλά μην ξεχνάμε και την, το πόσο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Η Europol παρακολούσε με μεγάλη προσοχή τις προσπάθειές μας και ξέρω ότι και στο μέλλον θα έχουμε την υποστήριξή της και θα έχουμε και τη δυνατότητα να βασιστούμε, να στηριχτούμε πάνω της, να, να γύρουμε πάνω της, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση. Κύριε Γέγκερ, έχετε την αίσθηση ότι ολόκληρες απικίες ε, καλαβρέζικες ε, εγκαταστάθηκαν στην ε, Γερμανία. Η κοινωνία των πολιτών πώς το βλέπει αυτό, ο γερμανικός πληθυσμός. Και βέβαια δεν θέλω να γενικεύσω εδώ, αλλά οι δικές μας διοκτικές και ερευνητικέ αρχές βλέπουν ένα ένα σχέδιο ας πούμε, των εγκληματικών οργανώσεων. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη οι εγκληματικές οργανώσεις. Ολόκληρες απικίες, ολόκληρα κλάν ε, μεταφέρονται, ας πούμε, μεταναστεύουν ας πούμε, στη Γερμανία. Ακόμα και Σικελοί, όχι μόνο οι Καλαβρέζοι μετα... μεταναστεύουν στην ε, Γερμανία και στηρίζονται σε φίλους, σε συγγενείς που έχουν ήδη εγκατασταθεί. Φτάνουν λοιπόν εκεί στη Γερμανία Ανοίγουν εστιατόρια, πιτσερίες και ασχολούνται με το εμπόριο. Εγώ όταν το είπα αυτό σε έναν ε, Γερμανό εισαγγελέα και σε έναν Γερμανό συνάδελφο πολιτικό, όταν του είπα τι σημαίνει ακριβώς αυτό, το γεγονός ότι τα συμφέροντα αυτής της ε, μαφίας μεταφέρθηκαν από την ε, Καλαβρία στη Γερμανία. Ήρθα σε επαφή με Ιταλούς ε, συναδέλφους, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με ομολόγους τους Γερμανούς και μου είπαν ότι είχαν τεράστια προβλήματα. Γιατί? Γιατί αν είχε καταστεί δυνατόν να συνεργαστούν αυτές οι αρχές ε, για να διερευνήσουν ε, μαφιόζικες σχέσεις, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Ο Γερμανός συνάδελφος όταν ρωτήθηκε είπε «Εμένα δεν ενδιαφέρουν που προέρχονται τα λεφτά. Το σημαντικό είναι αυτά τα λεφτά ε, είναι, το σημαντικό είναι τα, λεφτά αυτά που υπάρχουν είναι να χρησιμοποιούνται για να στηρίζουν τη γερμανική οικονομία. Βολικό είναι αυτό, ε. Αλλά δεν, δεν συνειδητοποιείται από αυτόν τον κύριο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη γερμανική οικονομία μπορεί η οικονομία σας, και αυτός ο κίνδυνος θα υλοποιηθεί σε λίγο, θα πέσει στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων. Μετά το Duisburg, τι αντίληψη έχει ο Γερμανός πολίτης. Θεωρούν ότι είναι ένα επεισόδιο έτσι μεμονωμένο το οποίο έληξε ή συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει πραγματικά πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, με αποφασιστικότητα με ανταλλαγή πληροφοριών, μα κυρίως με μέγιστη συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, με τις δικαστικές ερευνητικές αρχές δηλαδή των άλλων κρατών μελών. Όταν ε, είπατε ότι δεν σας καλύπτουν οι πολιτικοί, δηλαδή ότι τις ε, δράσεις της ε, γερμανικής αστυνομίας δεν τις στηρίζουν, δεν τις καλύπτουν οι πολιτικοί. Θα ήθελα να το καταλάβω λίγο αυτό καλύτερα. Γιατί θα ήθελα να συνεργαστώ μετά και να συζητήσω και να μεταφέρω τα όσα μου πείτε στους Γερμανούς συναδέλφους που απουσιάζουν από την αίθουσα. Τι κάλυψη θα θέλατε να σας δώσουν οι πολιτικοί, την οποία δεν σας δίνουν, τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γέγκερ για να μας απαντήσει και συνεχεία στον κύριο Ρότ και στον εισαγγελία Κρατέρη. Σας ευχαριστώ. Όπως είπε ο κύριος Ρότε, η γερμανική πολιτική ακόμα δεν έχει συλλάβει σε όλες τις, τις διαστάσεις την υπονόμευση της ε, πολιτικής και δημοκρατικής ζωής από τις εγκληματικές δραστηριότητες και δεν μιλώ μόνο για την τράγκεντα και η ρωσική μαφία ε, λόγω ε, και η ρωσική μαφία δραστηριοποιείται και η Γερμανία είναι ελκυστική για αυτούς και λόγω του δημοκρατικού πολιτεύματος και λόγω της ε, οικονομική της ευρωστίας. Η γερμανική πολιτική δεν είναι διατεθειμένη ακόμα να πει, όπως νομίζω ότι γίνεται στην Ιταλία, δεν αγοράζουν πλέον ε, υλικά, ε, είδη ε, πολυτελείας γιατί μετά τις 10.000 ευρώ πρέπει να δικαιολογήσουν πόθεν έσχον, τα χρήματα. Ενώ στη Γερμανία δεν σημαίνει αυτό. Έρχεται κάποιος Ιταλός και αγοράζει μια πιτσερία που κοστίζει 300.000 ευρώ και κανένας δεν ρωτά πόθεν έσχες τα χρήματα. Τώρα το εάν κάποια στιγμή αλλάξει η στάση αυτή της πολιτικής ε, τάξης είναι άγνωστο για μένα. Για την ώρα δεν το βλέπω πάντως. Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία θεωρώ ότι θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν από τα χρήματα της ε, Ιταλικής Μαφίας. Θα ήθελα να αρχίσω τώρα με την ερώτηση του Ευρωβουλευτού σας για το Ευρωπαϊκό FBI. Θα συμφωνήσω με τον Ισπανό Ευρωβουλευτή ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Έχουμε την Ευρωπόλ, η οποία είναι μια οργάνωση η οποία υποτίθεται ότι διασφαλίζει την πανευρωπαϊκή ανταλλαγή πληροφοριών και νομίζω ότι η αντιμετώπιση των εγκληματικών δραστηριοτήτων πρέπει να διεξάγεται στις χώρες προελεύσεως των εγκληματιών. Η Ιταλική αστυνομία ε, διώκει τις ε, ε, εγκληματικές δραστηριότητες των Ιταλών μαφιόζων σε όλη την Ευρώπη, όπου και αν συμβαίνουν. Ο Γκρατέρη εγκύπτει στα θέματα αυτά στην Καλαβρία. Εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη γλώσσα, γνωρίζουν τις παραδόσεις και δραστηριότητες Η γερμανική δικαιοσύνη δεν μπορεί με κανένα τρόπο να κατανοήσει πώς έχουν αναπτυχθεί αυτές οι εγκληματικές δομές επί δεκαετίες. Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν διάφοροι δράστες ή συνένοχοι. Εγώ μιλώ εκ μέρους του συνδέσμου των ε, Γερμανών αστυνομικών. Εγώ θα ήθελα να δω μια γερμανική, μια, ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Βεβαίως βήμα προς βήμα. Να γίνει πρώτα το βήμα η Ιταλία να δεχθεί τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Ανεξαρτήτως τώρα αν αντιστοιχούν στο Ιταλικό δίκαιο ή όχι. Να μπορούν να ε, περάσουν αυτά τα πράγματα, τα αποδεικτικά στοιχεία, ένα προς ένα στις ε, Ιταλικές ποινικέ διαδικασίες. Τώρα, για παράδειγμα, η Ρουμανία αποδεικτικα στοιχεια ενα προς ενα στις ιταλικες ποινικες αρμοδία για την δίωξη των διεθνών ποινικών πράξεων στην ε, ε, Ευρώπη και δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή η Βουλγαρία για τις δραστηριότητες των Βουλγάρων στην Ευρώπη και όλοι οι δράστες οι οποίοι προέρχονται από τη, ας μείνουμε γιατί στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στο Κόσοβο προέρχονται από εκεί όταν αυτοί δραστηριοποιούνται προσωρινά υπάρχουν και πολλοί ε, δράστες οι οποίοι ταξιδεύουν σήμερα στη Γερμανία, αύριο στη Γαλλία, μεθαύριο στην Ισπανία Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συλλεχθούν τα αποδεικτικά στοιχεία ανά χώρα και μετά να διαβιβαστούν στην ε, ε, Ρουμανία. Νομίζω ότι δεν μπορούν να απαλλαγούν οι χώρες αυτές από την ευθύνη, των, ε, από την ευθύνη να διώξουν τις εγκληματικές δράσεις των υπηκών τους. Δεν μπορούν να εξάγουν εγκληματίες. Η Λιθουανοί κλέφτες μηχανημάτων GPS οι οποίοι έχουν ειδικευθεί να κλέβουν τα μηχανήματα αυτά ε, ηλεκτρονικής πλοήγησης από πολυτελή γερμανικά αυτοκίνητα. Θα πρέπει να κάνουν τότε όπου, όπου διαπιστωθεί η εγκληματική αυτή δραστηριότητα να προβούν στη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και μετά να διαβιβαστούν στη Λιθουανία. Ε, ε, ε, εκεί πρέπει να γίνει η δίωξη. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα αυτοί οι Ευρωπαίοι εγκληματίες, το να διώκονται στις πατρίδες τους όπου και αν έχουν κάνει τις εγκληματικές δραστηριότητες. Και οι χώρες όπου έχουν γίνει οι εγκληματικές δραστηριότητες να μπορούν να στέλνουν στις σχετικές ποινικές διαδικασίες και παρατηρητές, ώστε να μην υπάρχουν, όπως είπαμε και προηγουμένως για διαφθορά, περιπτώσεις όπου αυτοί απαλλαγούν. Το ίδιο οι πορτοφολάδες από τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία που κλέβουν πορτοφόλια σήμερα στο Παρίσι, αύριο στην Αμβέρσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την Πανευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων για τους διεθνείς συγκληματίες και μετά πρέπει να ληφθεί μια απόφαση ποιος κάνει τις έρευνες σε βάρος αυτών των εγκληματιών. Αυτά πρέπει να τα κάνει μια κοινή οργάνωση, όχι όμως FBI. Πρέπει να έχουμε υπεύθυνου τους Ρουμάνους για τις εγκληματικές δράσεις των υπηκών τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Εμείς οι Γερμανοί αστυνομικοί θέλουμε να υπάρξουν joint investigation teams, μεικτές ομάδες που θα διεξάγουν ερευνός, μαζί δηλαδή με Ρουμάνους αστυνομικούς, με Βουλγάρους αστυνομικούς και μετά να αντιμετωπιστούν αυτές οι δομές, οι κλιματικές δομές, όπως κάνουν οι Ιταλοί με τη μαφία. Αυτό νομίζω ότι υπόσχεται κάποια επιτυχία. Εδώ στη Γερμανία διαπιστώνω ένα σημαντικό έλλειμμα με την έννοια ότι μεγάλος αριθμός των 16 ομοσπονδιακών κρατηδίων δεν υπάρχει καν εγκληματολογική εκπαίδευση. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ένας Ευρωπαίος αστυνομικό ειδικό στην δίωξη του εγκλήματο, ο οποίος να έχει ειδική εκπαίδευση, να γνωρίζει γλώσσες, να μπορεί να συνεργαστεί με άλλους Ευρωπαίους ε, αρμοδίους, να μπορεί ε, να χειριστεί ε, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων. Νομίζω ότι έχουμε εδώ δυνατότητες να βελτιώσουμε την απόδοσή μας ο Δανός Ευρωβουλευτής, οι αρνητικές πτυχές της ανταλλαγής δεδομένων. Εμείς δεν θεωρούμε ότι μετά από την σύμβαση του ΠΡΙΜ θα πρέπει κάθε αστυνομικός να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Μπορούν αυτά να διοχετευτούν σε συγκεκριμένους διάβλους. Μπορούν οι άνθρωποι που θα εργάζονται στις τράπεζες αυτές δεδομένων να ε, έχουν την ε, ε, υποχρέωση της εχεμήθειας δεν σημαίνει ότι ο τελευταίος αστυνομικός στο τελευταίο χωριό της Γερμανίας θα έχει πρόσβαση για, τους, ε, για όλους τους Ιταλούς μαφιόζους. Έχουμε στη Γερμανία φτιάξει κέντρα όπου συνέρχονται όλα τα δεδομένα σε ένα κέντρο και εκεί κάποια στιγμή ανάβει ένα λαμπάκι και λέει «Α, ποιον μπορεί να ενδιαφέρει η συγκεκριμένη πληροφορία». Αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η πρόσβαση για όλους τους αστυνομικούς σε όλα τα δεδομένα. Απλώς χρειάζεται καλύτερη συνεργασία έρχομαι σε αυτό που προτείνατε. Οι χώρες μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να συνεργαστούν με τρόπο ειλικρινή. Γι' αυτό και απευθύνω την έκκληση προς εσάς. Όσοι διαδίδουν ψεύδι να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Αυτό νομίζω το οφείλουμε και, στις, ε, και στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία και στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι η Γερμανία βρίσκεται στα νύχια της Ιταλικής μαφίας. Έχουμε μάλιστα λίγες διαδικασίες κατά της Ιταλικής μαφίας, διότι οι δραστηριότητες της προς τα έξω, όπως είπε και ο Γκρατέρη, δεν είναι τόσο ορατές. Και δεν έχουμε και τα απαραίτητο, το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσουμε να διώξουμε τέτοιες ε, ε, δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γέγερα. Δεν είπα ότι η Γερμανία βρίσκεται στα χέρια της μαφίας, αλλά ότι η γερμανική οικονομία είναι στο στόχαστρο της μαφίας, είτε είναι Ιταλικές είτε άλλες μαφίες διαφορετικής προέλευσης. Ο Γενικός Αγγελέας, ο κύριος ε, Κρατέλη, έχει το λόγο σε σχέση με το εμπόριο κοκαΐνης είναι πολύπλοκο το ζήτημα διότι τα εμπορευματοκιβώτια είναι το τελικό στάδιο της παράνομης διακίνησης της κοκαΐνης διότι το 80% πηγαίνει προς τη Δύση. Ένα 5 με 6% είναι ηρωίνη και τα άλλα είναι σύνθετα ναρκωτικά η Κολομβία, Βολιβία, Περού και Ουρουάη είναι άλλοι, ε, άλλοι διαφορετικές προελεύσεις, αλλά το 90% προέρχεται από την ε, Κολομβία. Το, τα Ηνωμένα Έθνη θεώρησαν ότι μπορούσαν να καταπολεμήσουν την ε, Κολομβία και τη διακίνηση ναρκωτικών στην Κολομβία. Πρόκειται για το 51ο έτος ε, ε, κράτος, με συγχωρείτε, των Ηνωμένων Εθνών. Και υπάρχουν ειδικέ ομάδες οι οποίες εργάζονται εξ ονόματος των Αμερικανών. Τους αγοράζουν, ε, τηλέφωνα, εξοπλισμό και ούτω καθεξής και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα αυτές οι ομάδες ε, κρούσης. Δεν πρόκειται για τους ε, μεγαλύτερους καταναλωτές κοκαίνης. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κοκαίνη προκαλεί μεγάλες ε, βλάβες στον εγκέφαλο και βλέπουμε ότι η κατανάλωση αυξάνεται η χρήση της κοκαίνης, ε, αυξάνεται και στην Ευρώπη, διότι δεν υπάρχει η σωστή εκπαίδευση. Τι κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ συμμετείχα στις ανακρίσεις του μεγαλύτερου εξαγωγέα κοκαίνης στον κόσμο ο οποίος είπε στις ανακριτικές αρχές ότι τα Ηνωμένα ε, Έθνη ε, έστελναν αεροπλάνα για να ψεκάσουν τις καλλιέργειες και εμείς στέλναμε αεροπλάνα που ψέκαζαν ε, με νερό τις καλλιέργειες. Δηλαδή, τι γινόταν, τους λέγαν ότι αν καλλιεργήσετε αραβόσιτο θα κερδίσετε 100. Ε, αν, αν καλλιεργήσετε κοκαίνη θα κερδίσετε 100, εάν, κερδί, καλλιεργήσετε αραβόσιτο θα κερδίσετε 60. Άρα οι καλλιεργητές ε, κοκαίνης άρχισαν να ξανακαλλιεργούν ε, κοκαίνη. Αν και ξέρουμε ότι μειώνεται η παραγωγή της ε, κοκαίνης σε αντίθεση με αυτό που μας δείχνει η κατάσταση στην Ευρώπη, όπου διακινείται η κοκαίνη. Πριν μιλήσουμε για τα εμπορευματοκιβώτια, θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι σε θέση να πούν στις πολυεθνικές τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή αυτοί που ε, δημιουργούν διάβλους επικοινωνίας όπως το Skype και άλλοι διάβλοι γιατί δεν πρέπει να ελέγξουν την κατάσταση. Δηλαδή τα κράτη της Ευρώπης ε, βρίσκονται υπό το ζυγό αυτών των πολυεθνικών που δημιουργούν διάβλους επικοινωνίας πάνω από τα κεφάλια μας, χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει πάνω από τα κεφάλια μας. Εμείς για να κάνουμε υποκλοπές στο Skype χρειαζόμαστε τέσσερα χρόνια να αποκωδικοποιήσουμε τα συστήματα. Δηλαδή όποιος εφήβρε το Skype θα πρέπει να μου δώσει τα κλειδιά αποκωδικοποίησης, αλλιώς να του βομβαρδίσω τους ε, δορυφόρους. Δηλαδή υπάρχει μία υπερστρωματοποίηση πάνω από τα κράτη και ο δυτικός κόσμος θα πρέπει να δράσει. Δεν ξέρουν τα κράτη τι συμβαίνει πάνω από τα κεφάλια μας μέσω των διάβλων επικοινωνίας. Αν μπορούσαμε λοιπόν να υποκλέψουμε εμείς τα νέα συστήματα επικοινωνίας, θα βρισκόμασταν πιο μπροστά από τις μαφίες. Σε σχέση με τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Ιταλία, θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο και με τις μεγαλύτερες εγγύησεις. Το πιο οικονομικό είναι γιατί χρειάζονται 4 ευρώ την ημέρα συν ΦΠΑ για να κάνετε υποκλοπή σε αυτό το τηλεφωνάκι που σας δείχνω. Και ξέρω τι γίνεται, δηλαδή εάν ο έμπορος κοκαΐνης είναι στην τουαλέτα ή πίνει τον καφέ του. Διαφορετικά θα πρέπει να γίνει παρακολούθηση από το Ρέτζο Καλάμπρια μέσω ε, μέχρι το Ρέτζο Εμίλια, το οποίο, χρειάζεται, το οποίο σημαίνει 2.000 ευρώ ημερησίως. Γιατί εγγυάται, τι εγγυάται, εγγυάται την φωνή, το τι λένε οι συνομιλούντες. Τι καλύτερη απόδειξη λοιπόν από αυτή της φωνής των συνομιλούντων. Όσο αφορά το εμπόριο κακοίνης, θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς κανόνες έτσι ώστε να μην συμφέρει κανείς να προβάλλει ε, παράνομες δραστηριότητες. Επειδή υπάρχει χαμηλότερη αξιοκρατία και δεν υπάρχουν πια αξίες, τότε μιλάμε γιατί μας αρμόζει καλύτερα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φυλάκισης, είμαι υπέρ των κανόνων. Θα πρέπει να είναι τέτοιοι κανόνες, ώστε να μην συμφέρει κανείς να προβεί σε παράνομες δραστηριότητες. Όταν λανθασμένα λέγεται ότι φοβούνται οι μαφιόζοι, ε, για τη δίμευση των αγαθών τους και όχι για τη φυλάκηση. αυτό το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Ναι, αυτό ισχύει, γιατί ο μαφιόζος βρίσκεται στη φυλακή 4-5 χρόνια που δεν είναι τίποτα στην μεγάλη του εγκληματική σταδιοδρομία. Εάν μιλάμε όμως για ποινές φυλάκισης 20 ετών και άνω, τότε θα τον απασχολούσε τον μαφιόζο και η φυλάκιση. Εσείς μιλήσατε για την Ελβετία και πολύ σωστά. Είναι μια μαύρη τρύπα η Ελβετία. Υπάρχουν πολλές ομάδες ντράγκετα. Ξέρετε τι υπάρχουν. Υπάρχουν, ε, ε υπάρχουν μάλλον ποινές της τάξης των 5 ετών. Γι' αυτό και υπάρχουν ομάδες της Ντράγκετα, της Καμόρα, της Κόζα Νόστρα, γιατί εκεί η φυλάκιση είναι πιο ήπια. Στην Ελβετία εννοώ. Εάν δεν διενεργηθούν έρευνες, πού ξέρουμε εάν δρά ή δεν δρά η Ντράγκετα. Ο Δανός ε, Ευρωβουλευτής ε, μίλησε για την Τράπεζα Δεδομένων. Μην ανησυχείτε. Ήμουνα και στην Κοπενχάγη και είδα ότι δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ορίσει καν το θέμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο δράμα και ξέρετε πόσο ξέπλυμα γίνεται στη Δανία. Τεράστιο. Όπως είπε και η κυρία Αλφάνο, θα πρέπει να υπάρξουν ε, αγαστές διεθνείς σχέσεις. Εγώ είμαι πολύ ευθύ στις παρεμβάσεις μου, γιατί μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Η καταπολέμηση της ε, μαφίας είναι σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό ε, δεν δέχομαι επικίνδυνες αποχρώσεις. Εάν μια χώρα αναλαμβάνει δεσμεύσεις δυνάμει της συνθήκης του Σέγγεν που χρησιμοποιούμε καθημερινά, δεν θα ήταν δυνατόν η Ολλανδία να μου πει ότι δεν μπορεί να κάνει υποκλοπές γιατί δεν έχει προσωπικό. Ή η Ισπανία να μου πει ότι δεν μπορεί να έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πάνω από δύο μήνες. Όταν μιλάμε για ε, τόνους, εκατοντάδες τόνων κοκαίνης που διακινούνται στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται 20 έρευνες ανά τον κόσμο και συνεργάζομαι με τα δικαστικά συστήματα 20 κρατών ανά τον κόσμο. Και μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συνεργάζομαι καλύτερα με Κολομβιανούς ή Βραζιλιάνους παρά με Ευρωπαίους. Ε, ως προς τη Μεγάλη Βρετανία θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν 42 ε, αστυνομικές ε, δυνάμεις ή ομάδες ή οργανισμοί. Υπάρχει αυτή η υπερβολική τυποποίηση στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο στην Αγγλία. Δηλαδή για μία λέξη, για, μία, για ένα κόμμα μας στέλνουν πίσω τις δικαστικές εντολές η κατάσταση βελτιώθηκε γιατί από την Βία έχουμε έναν υπεύθυνο ο οποίος μεταβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία στους διάφορους υπευθύνους και συνδιαλέγεται. Αλλά δεν είναι δυνατόν για ένα κόμμα να μου απορρίπτεται τη δικαστική εντολή και μετά να μου απαντάτε δύο μήνες μετά. Ξέρετε πότε απαντάει η Μεγάλη Βρετανία πρόσφατα διενεργήθηκε μία έρευνα όπου κατασχέσαμε 2.500 ε, ε, διαμερίσματα, σε 2.500 ε, διαμερίσματα και όταν είδαν ότι υπήρχε περίπτωση τρομοκρατικής δραστηριότητας μέσω Ήρα α, τότε τρελάθηκαν, μας τηλεφωνούσαν κάθε μέρα. Είχα την Scotland Yard στη διάθεσή μου, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Εγώ χρειάζομαι online ε, τα στοιχεία στη διάθεσή μου, ανεξάρτητα από την τυπολογία του εγκλήματος. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστούμε το Γενικό Ισαγγελέ. Τώρα ο κύριος Ρόφ έχει το λόγο. Κύριος σύντομα σχόλια. Καμιά φορά είναι ωραία να διακρίνεται, να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον τρόπο σκέπτεστε των πολιτικών από τους αστυνομικούς. Η οικονομική εγκληματικότητα, η διαφθορά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με νόμους. Άρα χρειάζεται να αναπτυχθεί μια κοινωνική συνείδηση. Χρειάζεται διαφάνεια, Χρειάζεται μια κουλτούρα της νομιμότητας, κάτι το οποίο ζητούν πολύ και στην Ιταλία. Εφόσον δεν γίνει αυτό, δεν σας εξυπηρετούν ούτε καλύτεροι νόμοι. Δεύτερο, η αστυνομία διακρίνει ανάμεσα στην κακή μαφία από τη μια μεριά και, από, και την πολιτική και την οικονομία από την άλλη μεριά. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχει πια αυτή η διάκριση τόσο πολύ και σίγουρα όχι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ θεωρώ όντως σημαντικό τον αγώνα κατά του ναρκωτικού, κατά της κοκαίνης, αλλά να μην λησμονούμε και την παγκόσμια οικονομική εγκληματικότητα, την παγκόσμια οικονομική βιομηχανία εντό εισαγωγικών. Η απειλή κατά τη δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών δεν είναι τόσο πολύ η κατάχρηση της κοκαίνης. Πιο πολύ είναι η Goldman και Sachs, να το πω έτσι κάπως απλά και συνθηματικά. Βρίσκω ότι εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη η σημασία των, η αρνητική δηλαδή σημασία των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι πάντοτε και αγώνας κατά εγκληματικών δομών. Εκεί καλείται να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια χώρα μέλος, η Βουλγαρία, που επικεφαλής της DANS, ένα είδος βουλγαρική, βουλγαρικού FBI, επικεφαλής διορίστηκε ένας ολιγάρχης με ένα ιδιαίτερα σκοτεινό παρελθόν αντέδρασαν και στην Σόφια υπήρξαν εντονότατες διαμαρτυρίες. Στο μεταξύ λοιπόν τον απέσυραν αυτόν. Αλλά φαίνεται καθαρά ποια είναι η επιρροή των κύκλων αυτών. Άλλο ένα παράδειγμα. Το Μαυροβούνιο είναι χώρα υποτίθεται θα ενταχθεί. Ο πρώην και νυν πρόεδρος Λουκάνοβιτς έχει εξαπατήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε φόρους ύψου 10 δισεκατομμυρίων. Είχε εκδοθεί Ιταλικό ένταλμα σύλληψη, αλλά δεν έγινε τίποτα γιατί όταν ήταν Πρωθυπουργό. Τώρα δεν τα συζητεί κανένα πλέον αυτά τα πράγματα. Όταν έχει τόσο πολύ αναμειχθεί το εγκληματικό με το πολιτικό επίπεδο, τι να σας πω, σα εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία ε, στην αντιμετώπιση και τον αγώνα κατά τη συνήθου ας πούμε, εγκληματική ε, δραστηριότητα. Ευχαριστώ κύριε Ρόθ. Ευχαριστώ τους ομιλητές αυτού του πάνελ για το πάθος με το οποίο εξέφρασαν τις απόψεις τους και ελπίζω και εύχομαι να ακουστείτε. Μπιλ, θες να πάρεις το λόγο τώρα? Δεν ξέρω αν θα φύγουν τώρα οι διερμηνείς ή αν έχουμε χρόνο να ξανακάνουμε ερωτήσεις στους ομιλητές. Ε, έχουμε χρόνο μέχρι τις 12.30, εδώ θα είναι, μέχρι τις 12.30. Έχουμε Μπιλ. φυσικά. Όμως, σας παρακαλώ σύντομα. Μόνο τα λεφτά έχουμε, Πρόεδρε. Έχουμε ακόμα ένα πάνελ ομιλητών. Δεν είναι το τελευταίο μας πάνελ αυτό. Έχουμε να μιλήσουμε με τους εκπροσώπους της ε, Υπηρεσίας Διώξης ε, Μαφίας. Κύριε Γέγκερ, κάθε αστυνομική αρχή κάθε κράτος μέλους πρέπει να ερευνά τους πολίτες της. Πώς συνεργάζεστε με τους ε, Ρουμάνους αστυνομικούς που θα μπορούσαν να πούμε να διώξουν Ρουμάνους εγκληματίες στη Φιλανδία. Θα μπορούσαν να το συλλάβουν. Οι μάρτυρες θα έπρεπε να πάνε πίσω στη Ρουμανία και ποιος θα πληρώσει για αυτή τη μεταφορά, ποιος θα δώσει διερμηνείς. Δεν νομίζω ότι δουλεύει το σύστημα. Αντίθετα με αυτά που είπε ο Ιταλός συναδελφός σας στα δεξιά, που λέει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, λεπτομέρειες και το τελευταίο κόμμα, ας πούμε, στην κάθε λέξη. Ε, τα 28 διαφορετικά συντάγματα. Κύριε Γέγκερ, δεν νομίζω ότι οι αστυνομικέ αρχέ πρέπει να είναι, του κάθε κράτους μέλου πρέπει να είναι υπεύθυνε μόνο για τους πολίτες του, για του πολίτε αυτού του κράτου η μόνη λύση είναι η ομοσπονδιακή λύση, όπου ξεπερνάμε τις πολλαπλές διαφορές και περνάμε σε μια ευρωπαϊκή λύση. Η περισσότερη Ευρώπη νομίζω ότι είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Ρώθες, που μιλήσατε στο τέλος, θαυμάσια τα είπατε, ε, εγκληματίες από το Μαυροβούνιο που δραστηριοποιούνται, ίσως σε 5-10 χρόνια ας πούμε, μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα αφήσουμε όλη αυτή την ευθύνη για τους ε, μαυροβούνιους εγκληματίες να κυνηγήσει τους μαυροβούνιους, να τους κυνηγήσει ανά την Ευρώπη η μαυροβουνιακή αστυνομία, μόνο, μόνη της, είναι δυνατόν. Πέστε μου, έχω άδικο. Ευχαριστώ, Μπίλ. Θα ήθελα οι απαντήσεις των ομιλητών να σταλούν γραπτός, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε το χρόνο που πρέπει στους ομιλητές του επόμενου πάνελ. Σας παρακαλώ να απαντήσετε γραπτός. Ε, girerà Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μα διαθέσατε και κυρίω για την παρουσίαση των ε, απόψεών σα Και τώρα καλά, καλό το Διευθυντή της ε, Υπηρεσίας Δίωξη Μαφίας, Αρτούντε Φιλίπε, τον ε, συνταγματάρχη της Υπηρεσίας Δίωξης Μαφίας του Παλέρμου, δύο άτομα που θα μας εξηγήσουν και οι δύο τις τελευταίες εξελίξεις στον αγώνα κατά πολέμηση της μαφίας, της υπηρεσίας αυτής. Και θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, τις τελευταίες εξελίξεις του αγώνα αυτού. Κάθε εισηγητής έχει στη διάθεσή του 20 λεφτά για την παρουσίαση της δουλειά του και μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν 20. 20 Θα δώσω το λόγο στον Αρτού Αντεφελίτσε, στο διευθυντή της υπηρεσίας αυτής διώξης μαφίας. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, και στον αστυνομικό διευθυντή θα ήθελα να εκφράσω τους χαιρετισμού μου. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να μιλήσω για να σας δώσω στοιχεία που γνωρίζω για τις τελευταίες εξελίξεις του αγώνα κατά της μαφίας και της δραστηριότητας της διεύθυνσης της οποίας προείσταμε. Μου ζητήθηκε να κάνω αυτή την παρουσίαση <clears throat> την 1η Νοεμβρίου του 2012. Ε, προσπαθώ να καταλάβω την απειλή που προέρχεται από τη μαφιόζικη και κλιματικότητα και φυσικά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις οικονομικές πτυχές του φαινομένου αυτού. Η οικονομική διάσταση του οργανωμένου εγκλήματος διαμακρών ε, μακρόν, μάλλον, είχε υποεκτιμηθεί. Δίναμε πάντα μεγαλύτερη σημασία στις ε, εκδηλώσεις βίας, που είναι κλασικές των εγκληματικών οργανώσεων, χαρακτηριστικές των εγκληματικών οργανώσεων, γιατί φυσικά αυτό προκαλούσαν ε, κοινωνικό συναγερμό. Και ασχολούμασταν βεβαίως με, τις, ε, με τα προβλήματα που δημιουργούσαν τα φαινόμενα αυτά στη δημόσια τάξη. Συν το χρόνο όμως, οι αρχές, οι, καταρχάς οι εθνικές αρχές, αλλά και οι διεθνείς ε, αρχές και φορείς, κατάλαβαν ότι και η οικονομική διάσταση της εγκλημα... του οργανωμένου εγκλήματος επηρεάζει τρομακτικά την τοπική οικονομία και καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες μέσω ενός ε, πολύ προηγμένου παράνομου δικτύ, διεθνούς ε, δικτύου όπου φέρνει σε επαφή τις διάφορες μαφίες μεταξύ τους. Η ανάλυση που έκανε η Υπηρεσία Δίωξης της Μαφίας επιβεβαιώνει τον κίνδυνο που προέρχεται από τις ομάδες αυτές ε, της μαφίας. Αυτές οι μαφίες έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης, πολύ καλής οργάνωσης και μπορούν να προσαρμόζονται στις διάφορες ενταφικές και κοινωνικές ε, πραγματικότητες. Ε, μερικές φορές αποποιούμενες και τα βασικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο ας πούμε της επικράτειας αυτής. Επιλέγουν μια στρατηγική έτσι, πιο χαμηλών τόνων, σχεδόν ε, γίνονται αόρατοι αν θέλετε. Συνεπώς, αυτό που με ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει είναι να ε, ελεγχθούν οι εγκληματικές δραστηριότητες και ο παράνομος ε, πλουτισμός. Μιλάμε για τεράστιο κεφάλαιο που απορρέει από παράνομο ε, εμπόριο που υπησέρχεται στον ιστό της οικονομίας και αποτελεί πραγματική απειλή για, την, ε, ε, για το ελεύθερο επιχειρήν, δημιουργώντας μεγάλες τρευλώσεις στην οικονομία. Αυτό το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο σε μία περίοδο μεγάλης ε, οικονομικοχρηματικής και οικονομικοπιστωτικής κρίσης. Άρα οι επιχειρήσεις της μαφίας έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι του ε, επιχειρηματία, ο οποίος είναι τίμιος, διότι διαθέτουν τεράστια κεφάλαια με μηδενικό κόστος. Έτσι, το οργανωμένο έγκλημα δραστηριοποιείται ολοένα και περισσότερο στην δημόσια ε, διοίκηση μέσα στα πλαίσια μιας συνενοχής με τον πολιτικό και διοικητικό τομέα. Με βάση τις εμπειρίες μας σε αυτό το τομέα, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η συνενοχή με τον πολιτικό και δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στα πλαίσια των δημόσιων προμηθειών όσον αφορά τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις, τη διάθεση των αποβλήτων και την απόκτηση αγαθών κάθε τύπου και την διαχείριση των υπηρεσιών. Η σύμιξη μεταξύ ε, οργανωμένου εγκλήματος πολιτικής και του κόσμου του επιχειρήν οδηγεί και σε σχέσεις στη δημόσια διοίκηση όπου υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό μέσα στα πλαίσια των ε, μεγάλων μόλ, των ε, τυχερών παιχνιδιών και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτική και δημόσια ζωή μέσω, ενό, μέσω ενός διάβλου επικοινωνίας. Το κοινό χαρακτηριστικό που διέπει τις εγκληματικές οργανώσεις που θέλουν να επηρεάσουν τη δημόσια διοίκηση αφορά τη διείσδυση ιδιαίτερα στον κοινωνικό ιστό. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το οργανωμένο έγκλημα πλήττει και την οικονομία, την νόμιμη οικονομία, καθώς και τη δημόσια διοίκηση. Μέσα στα πλαίσια αυτής της διείσδησης που επιτρέπει τον υπερβολικό πλουτισμό και γι' αυτό ακριβώς η Ιταλία έχει ένα ε, καινοτόμο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι πραγματικά ρηξικέλευτο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος για να μπορέσουμε να καλύψουμε το διτό στόχο καταπολέμησης της μαφίας και διασφάλισης της διαφάνειας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να διενεργούνται έρευνες, ε, δημεύσεις και ούτω καθεξής έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την πραγματική οικονομία καταπολεμώντας το κεφάλαιο αμφίβολης ε, προέλευσης. Επίσης, στον τομέα της, ε, της ε, δικαστικής συνεργασίας θα πρέπει να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε κοινοπραξία σε επίπεδο μαφίας που γίνεται δυνάμει του άρθρου 416α του ποινικού κώδικα της Ιταλίας ορίζοντας τους μηχανισμούς λειτουργίας και επιτρέποντας ε, την καταπολέμηση οποιοδήποτε αδικήματος και μέσα στα πλαίσια αποδεικτικών ε, στοιχείων. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο αφορά και την ε, εγκληματική δραστηριότητα που λειτουργεί εκτός Ιταλίας. Υπάρχει λοιπόν μία ενίσχυση και των ε, ποινών που επιβάλλονται στα, στις εγκληματικές αυτές δραστηριότητες, έτσι ώστε να ε, καθίσταται πιο εύκολη και η κατάσχεση ή δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Μίλαμε λοιπόν για δίμευση περιουσιακών στοιχείων για τους υπόδικους ή καταδικαστέντες για σοβαρά αδικήματα. Άρα μπορούν να κατασχεθούν και να δημευθούν αγαθά που δεν σχετίζονται άμεσα με ένα συγκεκριμένο αδίκημα, αλλά όταν αποτελούν, ε, υπάρχουν μάλλον αποδεικτικά στοιχεία ενός παράνομου πλουτισμού που δεν δικαιολογείται, δηλαδή που δεν υπάρχει σαφές πόθεν έσχες για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Η Ιταλία διαθέτει και έναν μηχανισμό κατάσκευσης και δίμευσης ελήψη ποινική καταδίκης μέσα στα πλαίσια ε, ενός καθεστώτος πρόληψης και καταπολέμησης της μαφίας που αποτελεί άξονα δραστηριοτήτων και έδωσε περίφημα αποτελέσματα. Υπ, αυτού, ε, αυτή την έννοια, ο Τζουζέπε Ντάγκατα, που είναι δίπλα μου και είναι υπεύθυνο του επιχειρησιακού κέντρου DIA του Παλέρμο, θα σας ε, μιλήσει για μία συγκεκριμένη περίπτωση πρόσφατης ε, κατάσχεσης ε, μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος όπως διενεργήθηκε πρόσφατα στη Σικελία. Σήμερα, μέσα στα πλαίσια των ε, μέτρων πρόληψης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κώδικα που ισχύει για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και που ε, εγκρίθηκε κατά τα τέλη του 2011. Έτσι μπορέσαμε να ενημερώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και να κινηθούμε και σε προληπτικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε την δραστηριότητα των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιαίτερα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, ο κώδικας αυτός ε, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος ε, φέρει και τεκμηρίωση, ασχολούνται και με την τεκμηρίωση των εγκληματικών δραστηριοτήτων και οτιδήποτε έχει σχέση με τη λειτουργία αυτή. Έχει ε, ιδρυθεί, έχει θεσμοθετηθεί και ένας νέος οργανισμός που είναι ο Εθνικός Οργανισμός διαχείρισης των κατασχεθέντων και δημευθέντων αγαθών που αποτελούν απόρρια εγκληματικής δραστηριότητας. Και αυτός ο κώδικας αποτελεί συνέχεια του νόμου ο οποίος εγκρίθηκε το 1991. Θα ήθελα να σας μιλήσω το, για το σύστημα, για το σκέλος της πρόληψης. Ε, σε αυτό το θέμα, με αυτό το θέμα ασχοληθήκατε και πριν. Πρόκειται για ένα εξοδικαστικό σύστημα το οποίο είναι, κινείται εκτός ποινικού πλαισίου και το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανεξάρτητα από τις διώξεις που θα γίνουν στη συνέχεια για να δούμε κατά πόσο ε, ο υποκείμενος ε, δίωξη έχει προβάλλει μία παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχουν και δραστηριότητες ε, κατά υποδίκων που δεν έχουν συνεργαστεί άμεσα με τη μαφία και έτσι μπορούμε να πλήξουμε και αυτό τον, αυτή την κρίζα ζώνη όπου δρούν πρόσωπα που αν και δεν συμμετέχουν, δεν είναι στρατολογημένα από τη μαφία, ε, δρούν αποφασιστικά και αποτελούν ένα σύνδεσμο δραστηριότητας για τις παράνομες οικονομικές ροές ε, μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας. Χρειαζόμαστε ενδείξεις λοιπόν, έτσι ώστε οι δικαστικές αρχές να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη αδικήματος. Επίσης, τα πλαίσια αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική μας ευθύνη έναντι αυτού του, αυτού του επικίνδυνου χαρακτήρα δραστηριότητας. Έτσι, οι εγκληματικές αυτές δραστηριότητες να μην μπορούν να διαθέτουν κεφάλαιο το οποίο απορρέει από παράνομες δραστηριότητες, ιδιαίτερα εμπόριο ναρκωτικών. Αποδίδοντας τα περιουσιακά αυτά στοιχεία στους δημόσιους φορείς. Αυτός ο κώδικας έχει χρησιμοποιηθεί και προληπτικά, επιτρέποντας να μπορέσουμε και σε περίπτωση θανάτου να ανακτήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία των εγκληματικών οργανώσεων, δηλαδή μέσα στα πλαίσια του κληρονομικού δικαίου να μην μπορέσουν να φτάσουν στους δικαιούχους κληρονόμους, εφόσον αποτελούν αντικείμενο αθέμητου πλουτισμού. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης ότι ο διευθυντής της ΔΙΑ έχει εξουσίες να μπορέσει να διαχειριστεί τα περιουσιακά στοιχεία και είναι και η μόνη αρχή, δημόσια αρχή που μπορεί να δράσει σε εθνικό επίπεδο. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και φαινόμενα διείσδυσης, ιδιαίτερα στους δημόσιους διαγωνισμούς και στα πλαίσια συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. Γι' αυτό όλες οι επιχειρήσεις που έρχονται σε επαφή με τις δημόσιες αρχές πριν συνάψουν σύμβαση θα πρέπει να έχουν δώσει επαρκή στοιχεία μη συνεργασίας με εγκληματικά στοιχεία. Και γι' αυτό θέλουμε να καταστήσουμε αυστηρότερο το πλαίσιο λειτουργίας έτσι ώστε κάθε νομαρχία να έχει έναν έλεγχο ε, προμηθείων για να ξέρουμε πώς ε, έχουν, πώς έχει και πώς μπορεί να τύχει διαχείρισης αυτό το λεγόμενο white list, έτσι ώστε να γίνονται και περιοδικοί έλεγχοι για να είμαστε σίγουροι ότι οι επιχειρήσεις αυτές που περιλαμβάνουν στο white list πραγματικά δεν έχουν προωθήσει ύποπτες δραστηριότητες. Μέσα στα πλαίσια του κανονιστικού αυτού πλαισίου για την πρόληψη υπάρχει και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος έτσι ώστε να προωθήσουμε ύποπτες κινήσεις μέσα στα πλαίσια του ξεπλήματος. Επίσης, η κεντρική μας τράπεζα θα πρέπει να δώσει στην ΔΙΑ όλες τις ε, τραπεζικές συναλλαγές που είναι ύποπτες για παράνομη δραστηριότητα. Για να δείτε καλύτερα το ρόλο αυτού του οργανισμού καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος της ΔΙΑ θα πρέπει να μιλήσω για την απαρχή της στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχε μία συγκεκριμένη ε, διάρθρωση όπου συμμετείχε η Δία μαζί με τις ε, δικαστικές αρχές και συνεργασία με τον ε, και συνεργασία με τη Δημόσια Εισαγγελία. Έτσι προωθούμε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες προληπτικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε σχέση με εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της μαφίας. Μιλάμε λοιπόν για μια συγκεκριμένη δράση που κινείται σε δύο επίπεδα. Προληπτικά και κατασταλτικά. Δηλαδή με βάση τη συνεργασία δικαστικών αρχών και αντίστοιχα δίμευση και κατάσχεση. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2012 έχουμε προβάλει 47 επιχειρήσεις με συγκεκριμένες ε, συλλήψεις. Συλλήψεις σε 215 διαμερίσματα. Μιλήσαμε για κατασχέσεις ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ. Σε σχέση με το προληπτικό σκέλος, έχει μεγάλη σημασία να προωθηθούν ερευνητικές δραστηριότητες για την καταστολή και τους διάβλους αυτούς που δημιουργούνται. Έτσι και με βάση και τις κατευθυντήριες ε, γραμμές των Ιταλικών αρχών προβαίνουμε στην συνεχή εποπτεία στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής ως προς συμμετοχή στους δημόσιους διαγωνισμούς και καταπολέμηση του αθέμητου κλουτισμού που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Με βάση λοιπόν αυτούς τους τομείς μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα εξής. Υπάρχει το κεντρικό παρατηρητήριο για τους ε, δημόσιους διαγωνισμούς και προμήθειες, όπου υπάρχει μία συνεχής εποπτεία συγκεντρωτικά και σε κεντρικό επίπεδο όλες οι, όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί και προμήθειες μέσα στα πλαίσια και ενόψη του, της ΕΞΠΟ του 2015 στο Μιλάνο. Αυτό αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς και μας ενδιαφέρουν οι ε, οδικές και σιδηροδρομικές, οι διαγωνισμοί που αφορούν τις οδικές αρτηρίες και τους σιδηροδρόμους μέσα στα πλαίσια των, της ανάληψης των δημόσιων αυτών έργων. Ε, βεβαίως επικαλούμε πάλι την ε, white list αυτή, αυτό τον ε, κατάλογο, όπου συμμετέχουν οι επιχειρήσεις υπεράνω πάσης υποψίας έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία εγκληματική διείσδυση ε, στους εμπλεκόμενους αυτούς φορείς. Πρόκειται για μια καθαρά ε, διοικητική δραστηριότητα, δηλαδή μια αυτόνομη ε, δραστηριότητα στα πλαίσια της ανάληψης και ανάθεσης ερευνών. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος για να αναλυφθεί η δράση. Υπάρχει και η πρόσβαση στις ε, διάφορες επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια αυτού του Interforce όπου συνεργάζονται οι, νομαρχια... οι νομαρχιακές αρχές. Θα ήθελα να μην επεκταθώ για να έχει χρόνο και ο επόμενος ομιλητής. Θα, θα ήθελα λοιπόν να σταθώ και σε ορισμένα στοιχεία τα οποία προαναφέρατε. Εμείς εκπροσωπούμε έναν οργανισμό στα πλαίσια της δημόσιας ασφάλειας που προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία εφήγησαν. Και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κεφάλαια που η μαφία προσπαθεί να επανεπενδύσει σε νόμιμες δραστηριότητες. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει η εξάλληψη αυτής της απειλής για να μην υπάρχει αυτή η διείσδυση στην νόμιμη οικονομία. Γι' αυτό και η Δία είναι ένας βασικός προμαχώνας για την καταπολέμηση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε στην εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου ενδοευρωπαϊκά και, τη συνεργασία, και να προωθήσουμε και τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Αρκετά χρόνια πριν, ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες, και όντας διευθυντής για τις εργασίες για τις ε, μελλοντικές, μελλοντική συμφωνία του Σέγγεν μέσα στα πλαίσια μία τράπεζας δεδομένων ε, της τράπεζας δεδομένων του NSIS είχαμε πολλές ελλείψεις και κενά αλλά επειδή υπήρχε καλή πρόθεση και καλή διαμεσολάβηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, φτάσαμε σε μία συμφωνία και αγαστή πραγματικά συνεργασία που έδωσε μεγάλους και σοβαρούς καρπούς. Είμαι λοιπόν ε, αισιόδοξο και πιστεύω ότι με μία ε, δραστήρια και αγαστή συνεργασία θα φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ντάγκατα, θα μας μιλήσει για μια συγκεκριμένη υπόθεση που τον απασχόλησε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ασχοληθώ με τις επιχειρησιακές ε, πτυχές της δράσης μας ε, κατά ε, παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών οργανώσεων. Θα μιλήσω για μία υπόθεση πολύ σημαντική που αφορούσε έναν ε, ε, ε, επιχειρηματία, τον Βίτον Ικάστρη, που δραστηριοποιείται στον τομέα της αιωλικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών. Το χρησιμοποίησε η Κόζα Νόστρα για να διεισδύσει στη νόμιμη οικονομία. τα περιουσιακά του στοιχεία καταρχάς τα κατασχέσαμε και συνεχεία τα δημεύσαμε θα, σταμα... θα σταθώ στην ε, ερευνητική μεθοδολογία, στο προφίλ του ατόμου αυτού του Νικάστρη και στα πιο σημαντικά αποτελέσματα που πέτυχε η Υπηρεσία Διοξυμαφίας του Παλέρμου και θα καταλήξω σε κάποια τελικά συμπεράσματα. Θα σταθώ στην προσωπικότητα του Νικάστρη, που είναι επιχειρηματίας από το Άλκαμο, που είναι μικρή γεωργική περιοχή στην προβίντσια του Τράπανη και που είναι ε, η πατρίδα του πιο διαβόητου φυγόδικου της μαφίας, του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Θα σταθώ λοιπόν στον Ικάστρη που τον εντοπίζουμε μέσα από την παρακολούθηση που έκανε μία ομάδα ε, με σκοπό να αναλύσει την εξέλιξη και τη δυναμική καθώς και την οικονομική διάσταση της Κόζα Νόστρα μέσα από μια συνεχή παρακολούθηση των ε, οικογενειών των μαφιόζων και των επενδύσεών του. Μετά από μια ανάλυση που κάναμε, ακολουθούν, ε, ακολούθησαν κάποιες έρευνες σε πιστοτικά ιδρύματα, σε χρηματοπιστωτικούς ενδιαμέσους και σε φορολογικές υπηρεσίες. Κάναμε αυτές τις επαφές για να εντοπίσουμε ε, όλους όσους διαχειρίζονται περιουσίες και αυτούς που δεν υποψιαζόμασταν και που κάνουν επενδύσεις ε, για, λογαριασμό, για ε, λογαριασμό της Κόζα Νόστρα. Από αυτή την ερευνητική δραστηριότητα Φτάσαμε λοιπόν στην, στην προσωπικότητα αυτή, στον Νικάστρη, που είναι επιχειρηματία στο τομέα της, των ανεώσιμων πηγών ενέργεια, ο οποίο ε, στο παρελθόν ε, είχε εμπλακεί σε πολλέ ποινικέ διοικέ ε, οικονομική και διοικητική φύσεω επίση ε, ε διαδικασίε. Από, αυτές, από αυτά όλα προέκυψαν σχέσει και επαφές του Νικάστρη με άλλου μαφιόζου, χωρίς όμως ε, ο ίδιος άμεσα ποτέ να έχει εμπλακεί σε έρευνες που αφορούσαν τη μαφία. Απλώς είχε επαφές με μαφιόσους. Όλα αυτά προκάλεσαν την, την προσοχή των αρχών ε, και εντοπίσαμε τις έρευνές μας στο άτομο αυτό. Σε άλλες παράλληλες έρευνες ε, διαπιστώσαμε ανάλογες συμπεριφορές διαφόρων άλλων επιχειρηματιών που έδειχναν ότι υπάρχει μια εγκύτητα, μια επαφή δική τους με εγκληματικές οργανώσεις. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε το προφίλ του Νικάστρη, μπορούμε να δούμε, ε, να πούμε τα εξής. Ότι ο Νικάστρη είναι 59 χρονών, ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή τη δεκαετία του 80, Καταρχάς δραστηριοποιήθηκε στον κοινωνικό γεωργικό τομέα ενό συνεταιρισμού και συνεχεία μαζί με τα αδέρφια του, τον Νικολό και τον Ρομπέρτο, ε, έγινε ηλεκτρολόγος και υδραυλικός, ε, έφτιαξε διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα της εγκατάστασης και της συντήρησης των κλιματιστικών. Μέχρι τελικά τη δεκαετία του 90 άρχισε να γίνεται πραγματικός επιχειρηματίας και να ασχολείται και με εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και τη δεκαετία 2000-2010 ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την εγκατάσταση εκμεταλλεύσεων για την, εναλλακτική, για την παραγωγή εναλλακτική ενέργεια και την παραγωγή συγγνώμη, ηλεκτρικής ενέργειας από εναλλακτικέ πηγέ, ε, χρησιμοποιώντας κυρίως το φωτοβολταϊκά και την ε, τα αιωλικά πάρκα. Και έγινε τελικά ένα είδος εργολάβου κλασικού έτσι, Ιταλού επιχειρηματία. Ο Νικάστρη ε, είναι αφιλεγόμενο άτομο, αήθης, ε, ικανός να κάνει οτιδήποτε, ε, το παίζει θύμα του συστήματος, που αναγκάστηκε ο καημένος να πληρώνει φακελάκια για να μπορέσει να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ε, ήδη από την δεκαετία του 1990 ήταν εμπλεγμένο σε μία έρευνα ε, διαφθοράς και παράνομης ύπαρξης ποσών. Ε, σε εκείνη την υπόθεση τότε, την δεκαετία του 90, δεν είχε κανένα κόλλημα να συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη. Ε, με τις έρευνες προσπαθήσαμε να απεικονίσουμε τις προσωπικές σχέσεις που, του ατόμου αυτού, ε, τις οικονομικές επαφές του και να δούμε πού μας οδηγούν όλες αυτές οι έρευνες. Καταλάβαμε ποια είναι η προσέγγιση του Νικάστρη. Ε, ο επιχειρηματής αυτός κατάφερε να φτιάξει πολλά αιωλικά πάρκα μέσω επαφών και συμφωνιών πολιτικών και μαφιόζων. Πολιτικών μαφιόζων και Νικάστρη. Ε, ήταν στο κέντρο ενός τριμερούς α, διεφθαρμένου συστήματος που έφερνε σε επαφή τρεις κόσμους. Το, τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες και τους μαφιόζους. Ο πολιτικός εξασφάλιζε στην ε, επιχείρηση τη διεκπαίρεση όλων των διοικητικών ενεργειών που ήταν απαραίτητες για την ε, δημιουργία των νεολικών ε, πάρκων και το, το αντιστάθμισμα ήταν ότι του υπόσχονταν φακελάκια, προμήθειες και τελικά του τα κατέβαλαν κιόλα. Ο μαφιόζος έδινε στην, στην επιχείρηση τη δυνατότητα να λειτουργήσει και στον πολιτικό να διαχειριστεί την υπόθεση και φυσικά με το αζημίωτο. Ο επιχειρηματίας ε, έκανε τη δουλειά του και έδινε δουλειά σε επιχειρήσεις με τη σειρά του που υποδείκνυαν ε, και ο μαφιόζος και ο πολιτικός. Αυτό το σύστημα που υλοποιήθηκε και απέδειξε την αξία του στην ε, Σικελία, το χρησιμοποίησε ο Νικάστρη και το εξήγηκε και στην Καλαβρία. Από τις έρευνες προέκυψαν σχέσεις με γνωστούς παράγοντες στην Τράγκετα, ε, στα κέντρα που έχουν πολύ ψηλή εγκληματικότητα της Καλαβρίας, Άφρικο, Πλάτη, Σαν Λούκα ε, με σκοπό την αγορά εδαφών ε, με σκοπό να υλοποιηθούν αιωλικά πάρκα. η μέθοδος ήταν πάντα η ίδια, επαφή με τους πολιτικούς οι οποίοι έδιναν την άδεια για να δημιουργηθούν αυτές οι επιχειρήσεις και με επαφή με τους τοπικούς μαφιώσους που εξασφάλιζαν τις την ήσυχη και ήρεμη διεξαγωγή των εργασιών. Και φυσικά και στους δύο, στους δύο αυτούς, πολιτικούς και μαφιόζους, έδινε φακελάκια. Από την έρευνα, ε, ο διευθυντής της ε, υπηρεσίας μας, ε, μετά την έρευνα μάλλον, υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο μια πρόταση για την διεξαγωγή προληπτικών μέτρων για τα άτομα και τις περιουσίες. Εν συνεχεία, οι αρμόδιοι δικαστές ε, δέχτηκαν ε, το κατηγορητήριο που βασιζόταν σε τρία βασικά στοιχεία, που ήταν η απλή ε, επικινδυνότητα του Νικάστρη που προέκυψε από έρευνες διοικητικής φύσεως και φορολογικής φύσεως. Η ειδική επικινδυνότητα που προέκυψε από μία σειρά σχέσεων και επαφών με στοιχεία της Κόζα Νόστρα και η οικονομική διαφορά Δηλαδή, η διαφορά ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που είχε και τις δηλώσεις που έκανε στις φορολογικές αρχές. Μετά από τις ε, προσπάθειες ε, κατάσχεσης ε, του δικαστηρίου, το Σεπτέμβριο του 2010 ξεκίνησε μια πραγματική διελκυστίνδα στη δικαιοσύνη και έγινε δίκη. Υπήρξε μάλιστα και η παρουσία ενός τρίτου δικαστή. Ε, το 2013 ε, στη δίκη ε, ολοκληρώθηκε η δίκη με την δίμευση των περιουσιακών στοιχείων. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ δημεύτηκαν και τέθηκε σε ειδική επιτήρηση ο Νικάστρη με υποχρέωση να διαμένει όντως στο Δήμο κατοικίας του. μετά από διάφορες ακροάσεις η Υπηρεσία Δίωξης Μαφίας συνέχισε και με την υποστήριξη του, συνέχισε να υποστηρίζει τον εισαγγελέα και προσπάθησε να, όλη αυτή η προσπάθεια είχε σκοπό να ενισχύσει τα αποδεκτικά στοιχεία εναντίον του Νικάστρη. Ε, όλα αυτά επιβεβαίωσαν ότι ήταν πραγματικά επικίνδυνο άτομο ο Νικάστρη. Με βάση... Επίσης, για πρώτη φορά ξεκίνησε μια σειρά ε, τηλεφωνικών υποκλοπών που έδειξαν την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο Νικάστρη για την οικονομική του δραστηριότητα. Από αυτή την τεχνική έρευνα επιβεβαιώθηκαν οι σχέσεις του Νικάστρη με τον πολιτικό κόσμο, με τον επιχειρηματικό κόσμο και με τον κόσμο της μαφίας. Από αυτές τις έρευνες, τις οποίες αξιοποιήθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο, μπορέσαμε να εμπλουτίσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Νικάστρη. Τελικά προέκυψε ότι ο Νικάστρη δεν είναι οργανικό τέλεχο, ε, δεν είναι πραγματικό μέλος της ε, Κοζανόστρα, αλλά είναι ένα επιχειρηματία που εποφελήθηκε από τη στήριξη της Κοζανόστρα την οικονομική δραστηριότητα και ε, έδωσε μια επίφαση νομιμότητας στην Κοζανόστρα και στις μαφιόζικες οικογένειε. Η μέθοδο αυτή του Νικάστρη δείχνουν το πώς εξελίσσεται η μαφία στην στις δραστηριότητές της, δηλαδή φέρνει σε επαφή τρεις κόσμους, τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες και τους μαφιούς, που κανονικά και θεωρητικά δεν θα έπρεπε να έχουν καμία σχέση. Ε, η εγκληματική οργάνωση αυτή έχει τεράστιο, τεράστιους πόρους, απίστευτο χρήμα για να προωθεί εγκληματικές δραστηριότητες ε, από λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, εκβιασμούς, διαχείριση τυχερών παιχνιδιών κτλ. Ε, και όλα αυτά τα χρήματα, η συνεχεία, τα ανακυκλώνει στην πραγματική οικονομία. Ε, με βάση λοιπόν διάφορα στοιχεία, με διάφορες, διάφορες ενδείξεις σοβαρές, συγκεκριμένες και διασταυρούμενες, μπόρεσε το δικαστήριο να προβεί στην κατάσχεση και δίμευση των περιουσιακών στοιχείων. Ε, επίσης αποδείχτηκε η διαφορά των οικονομικών στοιχείων ανάμεσα που δηλώνει ο Νικάστρο ότι έχει και που πραγματικά έχει. Ε, είχε περίπου 40 ε, ανώνυμες εταιρείε στον τομέα των ανεώσιμων πήγων ενέργειας, είχε περίπου 100 ακίνητα, είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα μεγάλου ε, κυβισμού, ένα καταμαράν, 70 ε, περίπου οικονομικές σχέσεις που όλες μας οδηγούσαν σε, σε άτομα τα οποία είναι υποέλεγχο και που διερευνούνται από τις αρχές. Ε, έχουμε διαπιστώσει στον τομέα της διανομής τροφίμων, σε σούπερ μάρκετ, στο τομέα του κατασκευαστικού τομέα, ε, στο κατασκευαστικό τομέα, στις ε, υπηρεσίες ε, στα λιμάνια και στην ανανεώσιμη ενέργεια ε, επενδύει λεφτά η, η μαφία. Επίσης, Ε, κάνουμε αυτή τη στιγμή έρευνε που θα, πιστεύουμε θα μα οδηγήσουν στην κατάσχεση περιφερειακών στοιχείων ύψου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία παράνομης ε, προέλευσης. Μετά από όλα αυτά κάνουμε διάφορε παρατηρήσει. Η Κοζανόστρα προσπαθεί να επενδύσει σε νέες οικονομικές δραστηριότητες. Ψάχνει πάντα να βρει αθώους, άτομα που δεν συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Ψάχνει επαγγελματίες, εμπόρους, ε, φοροτεχνικούς, ε, δικηγόρους, που ο καθένας με τον τομέα του και τις γνώσεις του κτλ. θα τη βοηθήσουν για να επενδύσει σε νέους οικονομικούς τομείς τα κεφάλαια τα οποία προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω κατά πόσο συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν, έχουν ερωτήσεις. Απλώς να ευχαριστήσω τους ε, δύο παρεμβαίνοντες, ε, Ντάγκατα και Φελίτσε, ε, για τον πολύ ζωντανό τρόπο έκθεσης του θέματος. Εγώ η Ιταλίδα από τη Σικελία και ιδιαίτερα από το Παλέρμο δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να τους ευχαριστήσω θερμά και εγώ θα είχα αρκετές ερωτήσεις γιατί και με τον δόκτωρα Ντεφελίτσε και με την Πρόεδρο μιλήσαμε για τις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχουμε χρόνο και δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Ε, θα ήθελα να κατανοήσω, να καταλάβω καλύτερα σε σχέση με την ε, εμπειρία σας στη ΣΥΠΑ, όπου υπάρχουν μυριάδες ερευνητικές ε, επιτροπές και σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει στην Ευρώπη, ποια θα πρέπει να είναι η θέση μας εδώ στην Ευρώπη σε σχέση με τον συντονισμό αυτών των, των αστυνομικών αρχών, των υπηρεσιών, πληροφοριών, τι θα μπορούσαμε να προσλάβουμε από το αμερικανικό μοντέλο Μία απάντηση θα ήθελα να σας πω. Η Δία είναι η Ιταλική απάντηση σε ένα θέμα που 20 χρόνια πριν μας απασχολούσε μόνο στην Ιταλία και που τώρα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, διότι ε, συνειδητοποίησαμε όλοι ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ένα σικελικό ή ιταλικό φαινόμενο, αλλά ευρωπαϊκό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η γενικότερη συνειδητοποίηση. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου. Να προωθήσουμε αυτή την ερευνητική διαδικασία επιτάπητος για τα καθημών γιατί αυτό μου ε, ε, μας ενδιέφερε ήταν να πάρουμε πληροφορίες και από το Ινστιτούτο Max ε, Planck στο Φράιμπουργκ για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δικά μας εντάλματα συλλήψεως και σε άλλες χώρες με βάση τις τράπεζες δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί φυσικά οι ένομες τάξεις ε, δεν συμπίπτουν οι εσωτερικές ένομες τάξεις και γι' αυτό νομίζω ότι η, το, Ιταλική αυτή ε, εμπειρία θα μπορέσει να αποτελέσει εφαλτήριο για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους ε, διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνταγματάρχη Ντάγκατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθημερινή δέσμευσή σας, για την προσπάθεια να ανταποκριθείτε και στο έργο σας γενικότερα, γιατί ξέρετε ότι και εμείς ασχολούμαστε με τη δίμευση κατάσχεση ε, αγαθών. Ε, που απορρέουν από εγκληματικές δραστηριότητες. Ε, μας ενδιαφέρει λοιπόν και η δική σας συνεισφορά διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που μετρά καθημερινά είναι τα αποτελέσματα. Πρόκειται λοιπόν για αυτά αποτελέσματα ύψης της σημασίας. Ευχαριστώ τον Διευθυντή Ντεφελίτσε για τη δραστηριότητά του μέσα στα πλαίσια της ΔΙΑ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω το θαυμασμό μου για αυτή την υποδομή η οποία προβλέπει 3.000 ε, θέσεις αλλά διαθέτει μόνο το ίμιση. Παρόλα αυτά όμως φέρει σε πέρας αυτή την εξαιρετική εργασία που καθημερινά δίνουν αυτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, διακόπτουμε και θα τα ξαναπούμε στις 3 η ώρα με την έκθεση του κυρίου Γιακολίνου.